Θα ήθελα επ' ευκαιρίας να σας ευχαριστήσω θερμά για την ολοκλήρωση των πολυσύντατων αυτών διαπραγματεύσεων, όχι μόνο για τέτοια θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα ομολογουμένως, αλλά και για τα θέματα νομίμης μετανάστευσης που εντάσσονται στην Λισαβόνα, για τα οποία προφανώς είναι πάρα πολύ ευαίσθητα θέματα στο τρέχον συγκείμενο. Άρα τεχνικός πώ ήταν πάρα πολύ αποδοτικοί και νομίζω ότι κατανοήσατε όλες τις πτυχές του θέματος. Αυτό θα βοηθήσει τους, τον κόσμο που επηρεάζεται από την νομοθεσία αυτή. Και θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους, τους υπόλοιπους συναδέλφους και όλους όσους ε, συμμετείχαν στο έργο αυτό. Ευχαριστώ. So, if there were, I should have asked if there were any other ρωτήσω από πριν αν υπήρχαν άλλα σχόλια, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Επειδή έχουμε κάποιες αλλαγές και στην ημερήσια διάταξη, να περάσουμε στο σημείο 6. Μια ενιαία θεώρηση, τύπος ε, θεώρησης. Η Σιλβί Βον Κάφμαν είναι η συγγήτρια. Έχουμε αυτό το αυτοκόλλητο θεώρησης ε, το οποίο ε, κυκλοφορεί εδώ και 20 χρόνια. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα νέο κοινό πρότυπο με κοινά χαρακτηριστικά, εξαφανισμένα χαρακτηριστικά ασφαλεία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κυρία Συγγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το περιγράψατε πριν από λίγο. Εδώ και πολύ καιρό έχουμε ένα ε, ενιαίο αυτοκόλλητο για τις θεωρήσεις, αλλά διαπιστώθηκε δυστυχώς ότι υπήρχαν και παραποίησεις ε, του αυτοκόλλητου αυτού. Ως εκ τούτου λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προτείνει να υπάρξει ένα νέο τέτοιο αυτοκόλλητο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, για να υπάρχει ένα ασφαλές ε, αυτοκόλλητο που να μην αντιγράφεται και επίσης ε, αυτό το αυτοκόλλητο να αποτελεί τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ε, αναπτύχθηκε λοιπόν τέχνικα μέσω συμβουλών των ειδικών αυτό το αυτοκόλλητο. Προτείνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και εγώ ω εισηγήτρια ότι είμαι πεπισμένη ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι δεν χρειάζεται οποιαδήποτε τροποποίηση στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έτσι δεν έχω τίποτα άλλο να σα πω. Ε, σύντομα και απλά τα πράγματα για την έκθεσή μου. Μέχρι 11 Δεκεμβρίου νομίζω ότι είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και αν οι συνάδελφοι επιθυμούν να καταθέσουν τροπολογίες Α το κάνουν, αλλά θα προτιμούσα να ακολουθήσουν την πρότασή μου, να σας πω την αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δύο σκιώδεις έχουν ζητήσει το λόγο. Κύριος Βός από το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ μιλάω εξ ονόματος του Πετρή Σάβαμα, ο οποίος μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία Κάουφμαν για την καλή και γοργή εργασία σας. Κατανοώ πόσο κατεπήγον είναι το θέμα αυτό και πόσο ε, έχει να κάνει και με θέματα ασφαλείας αυτή, αυτός ο εξυγχρονισμός του αυτοκόλλητου για να μην ε, μπορεί να αντιγραφεί. Άρα είμαστε υπέρ μιας γρήγορης διαδικασίας νομοθεσίας και λοιπόν ο συνάδελφος δεν πιστεύει ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκιώτες από τους φιλελεύθερους, ο κύριος Ντεπρέ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, με την οποία συμφωνώ επί της επιχειρηματολογίας και επί των συμπερασμάτων. Δεν θα υποβάλουμε λοιπόν τροπολογίες. Μόνο ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από καθαρά τεχνολογικής σκοπιάς. Αυτό το νέο μοντέλο θεώρησης αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ε, τη δυνατότητα να υπάρχουν και τα ευφυή σύνορα και έτσι να έχουμε και ε, αυτοματοποιημένη Θα ήθελα να ακούσω την απάντηση της Κομισιόν επί τούτου. Ναι, να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, απαντήστε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και την ερώτηση την οποία θέσατε να απαντήσω εν συντομία. Αυτέ οι ετικέτες, αυτά τα αυτοκόλλητα θεωρήσεων διαβάζονται από μηχανήματα. Αυτό τι σημαίνει ότι αυτή η ζώνη η οποία περνάει από το μηχάνημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές ICAO συμπεριλαμβάνεται σε κάθε ε, διαβατήριο και μπορεί λοιπόν αυτόματα να αναγνωστεί από τις μηχανές ε, που υπάρχουν σε κάθε σταθμό. Άρα βάζουμε λοιπόν ε, τα, στα μηχανήματα το διαβατήριο το οποίο και διαβάζεται. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι υπάρχει ένα τσίπ το οποίο συμπεριλαμβάνει βιομετρικές πληροφορίες και το οποίο δεν χρειάζεται επαφή με το μηχάνημα. Αυτά λοιπόν δεν περιλαμβάνονται στη θεώρηση αυτά τα στοιχεία, αυτές οι πληροφορίες, αλλά έχουμε το σύστημα πληροφοριών θεωρήσεων, όπου με την αριθμό του αυτοκόλλητου της θεωρήσεων μπορεί κανείς να κάνει αναζήτηση. Άρα υπάρχει σύνδεση των βιομητρικών πληροφοριών στο σύστημα πληροφοριών θεωρήσεων που συνδέεται με τον αριθμό του αυτοκόλλητου της ετικέτας της θεώρησης. Ελπίζω έτσι να απαντώ στην ερώτησή σας. It does. Okay. δεν ξέρω αν έχεις ε, περαιτέρω σχόλια. Μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι μπορείτε να υποβάλλετε Σε Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο σημείο 7. για την άνοιξη τη αυτοματοποιημένη συντελέχη δεδομένων σχετικά με τι άδειε κυκλοφορία οχημάτων στη Λετωνία παρουσίαση από την Προεδρία του Συμβουλίου και παρουσίαση της έκθεσης, του σχεδίου έκθεσης. Το Συμβούλιο λοιπόν θα μας παρουσιάσει το σχέδιο απόφασης ε, για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων, τη λεγόμενη απόφαση PRIM, σε ό,τι αφορά τη Λετωνία. Η κυρία Ένστ δεν είναι εδώ. Α, μια μικρή αλλαγή στην αλήθεια. Κυρία Πλάιν, θα μας παρουσιάσει το σχέδιο απόφασης ε, του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων, τη λεγόμενη απόφαση Παρακαλώ. Ευχαριστώ, τσέπμα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω συντομία την έκθεση σε ό,τι αφορά, μάλλον την ε, απόφαση του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τι κυκλοφορίε στη Λετωνία. Έχουμε υλοποιήσει γενικέ διατάξει ε, για την προστασία δεδομένων που εγγράφονται ε, την 615 απόφαση του 2008. Βάσει τη απόφαση πριν λοιπόν είναι απαραίτητη προπόθεση η έναρξη τη αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων εν γέννη και ειδικότερα ανταλλαγή δεδομένων σε σχέση με τα ανταλλακτικά αποτυπώματα. Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου στι 11 Νοεμβρίου του 2015 υπέβαλε την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Λετωνίας προς το Κοινοβούλιο προς έγκριση. Και έτσι ζητήσαμε και το Κοινοβούλιο να μας δώσει την ομοδότησή του εντός ε, τριών μηνών. Για να ενισχύσουμε την, ε, ε, την διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία καταπολεμώντας και την τρομοκρατία και το ε, διασυνοριακό έγκλημα, το Συμβούλιο θα ήταν ευγνώμων αν θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να υποβάλει τη γνωμοδότησή του το συντομότερο δυνατών. Και αυτό θα μας επέτρεπε να προχωρήσουμε στο τελικό βήμα υλοποίηση αυτών των εκκλησικών αποφάσεων του Συμβουλίου χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ. So, I think... Εδώ οι συντονιστέ αποφάσισαν βάσει του κανόνα να πάει η έκθεση στην ΕΓΚΟΕ. Θα ενημερώσουμε ότι δεν είναι εδώ η κυρία Ένστη για να απαντήσει, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος από την ΚΟΕ. Εάν όχι, να πω ότι το χρονοδιάγραμμα είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, γιατί έχουμε τρεις μήνες από το Συμβούλιο, επομένω ε, οι τροπολογίες θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 8 Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι. Αυτά για αυτό το σημείο. Επειδή δεν είναι εδώ και η κυρία Ένστ. Αλλά σίγουρα στο μέλλον ε, θα έχει τη δυνατότητα να πάρει το λόγο. Ωραία. we to point 8, uh, which is communication. Πάμε στο σημείο 8, ανακοίνωση της Επιτροπής ε, προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΕΕΠΑ υπό την οδηγία 9546 μετά την απόφαση του δικαστηρίου ε, στην υπόθεση ΣΡΕΜΣ. Sorry, colleagues, it's one of those afternoons. Yet. So, Okay. Λοιπόν, συνάδελφοι, επόμενο σημείο κανονικά είχαμε την παρουσίαση Τι περιμένουμε την Κομισιόν. Περιμένουμε λοιπόν να έρθει ο κύριος Φωνσέκα Μορίγιο, ο οποίος θα είναι εδώ σε 10 λεπτά και μου λένε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα 10 λεπτών, ζητώ συγγνώμη, ε, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα. 10 λεπτά, όχι αργότερα, θα είναι εδώ εντός 10 λεπτών και να συνεχίσουμε μετά. So please be back. Παρακαλώ λοιπόν να επιστρέψετε σε 10 λεπτά. How am I doing today? <clears throat> Συνάδελφοι, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Κύριος Μωρίγιο είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε την συζήτηση και την παρουσίαση της Κομισιόν για την ανακοίνωσή της του Νοεμβρίου. Κατανοώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το ζήτημα. Βεβαίως είναι τόσο φορτωμένη μέσα διάταξη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και μετά την ε, απόφαση ΣΕΜ έχουν υπάρξει και πολλέ άλλε εξελίξει. Όμω έχουμε προσχεθεί να κάνουμε μία λεπτομερή συζήτηση ε, για την υπόθεση αυτή και παρουσίαση τη ανακοίνωση τη 6 η Νοεμβρίου. Θέλω λοιπόν και οι σκιώδει να πάρουν το λόγο και να γίνει και μια ευρύτερη συζήτηση. Έχουμε χρόνο και γι' αυτό. Ο κύριος Μωρίγιο, από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μα κάνει την αρχική παρουσίαση με τα κύρια σημεία τη ανακοίνωση ε, του Νοεμβρίου. Και μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Λυπάμαι για την καθυστέρηση. Υπήρξε παρεξήγηση. Νόμιζα ότι 4 παρα 10 θα συζητιόταν το δικό μου ζήτημα, αλλά συμβαίνουν αυτά. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Όπως ξέρετε, πριν από 8 εβδομάδες, ε, το δικαστήριο Ε, κατέστησε άκυρη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό επιβεβαιώνει την σημασία των προσωπικών δεδομένων και της προστασίας τους όπως αυτή έχει καθιερωθεί και από τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπάρχει μια νομική, ένα συγκεκριμένο μήνυμα σε αυτή την απόφαση του δικαστηρίου. Τα προσωπικά δεδομένα όχι μόνο θα πρέπει να προστατεύονται κατά την επεξεργασία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό ισχύει και όταν τα δεδομένα διαβιβάζονται και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση. Με άλλα λόγια, το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων συνοδεύει τα δεδομένα, όπου και αν πάνε αυτά. Λαμβάνοντα αυτό υπόψη, θεωρούμε ότι ένα ανανεωμένος ασφαλή λιμένας είναι καλύτερη λύση και για την προστασία των δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και για την οικονομία μας η οποία εξαρτάται και είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τις ροές δεδομένων ε, από και προς της ΕΠΑ. Γι' αυτό θα πρέπει ε, να ενισχύσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις μας με την Αμερικανική Διοίκηση μετά τη δικαστική απόφαση και τώρα έχουμε σαφείς δείκτες τους οποίους θα αναφέρω στη συνέχεια. Η ακύρωση του Safe Harbor μας έχει κλείσει μια μεγάλη ε, δίωδο που αξιοποιούσαν ε, χιλιάδες επιχειρήσεων και έχει οδηγήσει σε μια τεράστια σύγχυση και αβεβαιότητα. Πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί που εκπροσωπούν επιχειρήσεις ε, ήρθαν σε επαφή μαζί μας μετά την δικαστική αυτή απόφαση, αλλά και εμείς από μόνοι μας ήρθαμε σε επαφή με πολλές επιχειρήσεις και οι περισσότεροι ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδώσει ασφάλεια δικαίου. Βεβαίω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ούτε ο μόνος, ούτε καν ο πιο σημαντικός παίκτη σε, αυτό το παιχνίδι. Η εποπτεία της προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πρώτον και κύριον ρόλος και αρμοδιότητα των εθνικών αρχών προστασία δεδομένων. Αυτό είναι και ένα από τα κύρια σημεία της δικαστικής απόφασης του ΕΜΣ. Κατανοείται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ιδιαίτερη επιφύλαξη ή μάλλον με ιδιαίτερα προσοχή προσπάθησε ε, να ακολουθήσει ακριβώς αυτές τις ε, προϋποθέσεις. Σε ό,τι αφορά τις ε, αρχές προστασία δεδομένων και η Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασία Δεδομένων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται στενά μεταξύ τους σε όλα αυτά τα στοιχεία και θέματα που αφορούν τα, ε, την προστασία δεδομένων, όπω γίνεται και στην ε, ομάδα, τη λεγόμενη ομάδα του άρθρου 29. Η ομάδα ε, εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία ήδη ζήτησε από όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να βρουν μια λύση με τι Αμερικανικέ Αρχές ε, μεταξύ άλλων και με μια νέα συμφωνία για έναν ανανεωμένο ασφαλή λιμένα. Ταυτόχρονα η ομάδα εργασία θα εξακολουθήσει να αναλύει ε, τον αντίκτυπο της ε, δικαστικής απόφασης ΡΕΜΣ, όμως αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιούν τις συνήθεις συμβατικές ρήτρες τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2016. Αυτό είναι μια συγκεκριμένη διευκρίνηση γιατί ε, δίνει αυτή την απαραίτητη ασφαλεία δικαίωση επιχειρήσει. Η ανακοίνωση της Κομισιόν προ το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη διαβίβαση δεδομένων ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς ε, της ΕΠΑ μετά την δικαστική αυτή απόφαση συνδέεται και με την δήλωση της ομάδας εργασίας. Δεν πρόκειται για νομοθετικό κείμενο η πρόθεσή μας δεν ήταν να νομοθετήσουμε, αλλά να διευκρινίσουμε τα ήδη ισχύοντα. Βασιζόμενοι σε προηγούμενα έγγραφα ε, κατευθυντήριων γραμμών που έχει εκδώσει η ομάδα εργασίας τα τελευταία χρόνια. Ελπίζουμε το αποτέλεσμα να είναι ένα συνεκτικό και εύληπτο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά μια επισκόπηση των επι, επιμέρους ε, μέρων μέσων μάλλον που έχουν όλη τη διάθεσή τους σε ό,τι αφορά ε, και την οδηγία προς τους δεδομένων. Οι δύο κύριες βάσεις είναι οι εξής. Οι συνήθει σημαντικέ ε, ρήτρε μεταξύ επιχειρήσεων ε, και Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτη χώρα, για παράδειγμα η ΕΠΑ, και εδώ διευκρινίζονται υποχρεώσει ότι αφορά την προστασία δεδομένων που θα πρέπει να τηρούνται και από την από αυτούς που εξάγουν δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την επιχείρηση υποδοχής, ο λεγόμενος Data Importer. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει τέσσερα σύνολα τέτοιων ρητρών που ε, χρησιμοποιούνται ευρέως από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δεύτερον, ε, δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες σε ό,τι αφορά τις ε, διαβιβάσεις δεδομένων στο πλαίσιο μιας πολυεθνικής. Όπως και η πρώτη κατηγορία και αυτοί οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες παρέχουν δικλείδες ασφαλείας ότι φορτή τους δεδομένων, αλλά ε, εγκρίνονται και από τις εθνικές αρχές τους δεδομένων. Επιπλέον, έχουμε και τους ευρωπαϊκούς κανόνες τους δεδομένων και έτσι υπάρχουν ε, ε, κάποιες δικλείδες ασφαλείας και χέγγια για την ασφαλή ε, διαβίβαση δεδομένων. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία. Τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σύναυση μιας σύμβασης. Δεύτερον, ε, οι διαβιβάσεις που είναι απαραίτητες για την άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Τρίτη προϋπόθεση, ότι η υπερασπιση νομικων αξιωσεων τριτη προποθεση βασίζεται και στην πλήρη συγκατάθεση του ε, ενδιαφερομένου. Και γενικά υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις ε, για αυτή τη διαβίβαση, όμως είναι σαφές και το καταστήσαμε κι εμείς ε, σαφές στην ανακοίνωσή μας, ότι όλες αυτές οι επιλογές είναι πιο περιοριστικές, ευαχθείς και δίνουν λιγότερη ασφάλεια δικαίου από ε, μια πραγματική απόφαση επάρκειας. Αυτά τα μέτρα τη φύση τους είναι έκτακτα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βασίζονται στην συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για να κάνουν τη διαβίβαση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει και ο ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται για τους πιθανούς κινδύνους που ενδεχομένως να ενέχει η διαβίβαση των δεδομένων του σε τρίτη χώρα. Καθώ η ανεπάρκεια συγκεκριμένων δεδομένων μπορεί να αποτελέσει και έλλειψη στην κατάσταση. Αυτό αποτελεί σημαντικό άχθο ε, για τι επιχειρήσει που θέλουν να διαβιβάσουν δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ε, γνωρίζετε, οι επιχειρήσει αντιμετωπίζουν σημαντικού περιορισμού όταν ε, βασίζονται σε εναλλακτικά μέσα διαβίβαση. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι χρειαζόμαστε ένα νέο, ενδυναμωμένο, πιο ισχυρό πλαίσιο υπερατλαντικών, διατλαντικών ε, ε, διαβιβάσεων προσωπικών δεδομένων που θα αντικαταστήσει τον παλιό Safe Harbor. Η συμφωνία Safe Harbor και οι διαπραγματεύσει μας με, την, με τη ΣΥΠΑ θα πρέπει να συνεχιστούν. Και αποτελεί και παραμένει βασική προτεραιότητα. Από τότε που η επίτροπο Γιουρόβα σας ε, ενημέρωσε στι 26 ε, Δεκεμβρίου, Οκτωβρίου, υπήρξαν πολλοί γύροι συζητήσεων με τις ΗΠΑ, ε, κυρίω σε τεχνικό επίπεδο. Και η ίδια Επίτροπος μετέβη στην Ουάσιγκτον στα μέσα Νοεμβρίου για να προχωρήσουν οι συζητήσεις για τον ασφαλή λιμένα. Και όταν ήταν στη Ουάσιγκτον είχε και πολλέ διμερεί επαφέ, με πολλά, πολλούς εκπροσώπους της Μεκανικής Διοίκησης, από το Υπουργείο Εμπορίου, ε, αλλά και από, τις, ε, από την Υπηρεσία Πληροφοριών. Συζήτησε το θέμα και με το Λευκό Οίκο, το State Department, αλλά και πολλά μέλη του Κογκρέσου. Επιπλέον, η Επίτροπος συμμετείχε σε μια σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Τρία είναι τα μηνύματα που ήθελα να προστείλει. Ενώ θέλουμε να υπάρξει και μια νέα απόφαση μετά το Safe Harbor, ο πύχης έχει δεχθεί υψηλά. Γιατί θα πρέπει να συμμορφωθούμε και με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το δικαστήριο στη δικαστική αυτή απόφαση. Δεν είμαστε στο σενάριο business as usual. Χρειαζόμαστε μια νέα συμφωνία που να είναι αλεξίσφαιρη. Γι' αυτό, Πρόεδρος Άντσιπ, τόνισε το αυτό ακριβώς το στοιχείο ε, στην ανακοίνωση και παραμένει ε, βασική μας αρχή. Πρέπει να βασιστούμε και στις ε, προηγούμενες εργασίες που είχαν γίνει με τη Αμερικανική πλευρά όταν είχαμε τις 13 συστάσεις πριν από δύο χρόνια. Οποιαδήποτε νέα συμφωνία θα πρέπει να είναι σταθερή και ασφαλής. Τέλος, εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να προχωρήσουμε στη σύνδεση νέας συμφωνίας. Όμως, πρέπει αυτό να έρθει και από τις δύο πλευρές. Και η αμερικανική πλευρά, η εταίροι μας, θα πρέπει να ε, εργαστούν μαζί μας ε, επικοδομητικά. Γιατί το σημαντικό δεν είναι τι λέμε στις εφημερίδες, αλλά τι ακριβώς λέμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Για τα τέλη Ιανουαρίου 2016 έχουμε θέσει μια προθεσμία να καταλήξουμε σε νέα συμφωνία. Όμως, ε, παρότι είναι δύσκολο, θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν και οι δύο πλευρές, και δηλαδή οι Αμερικανοί, το επιθυμούν πραγματικά. Μέχρι τώρα οι συζητήσει μας επικεντρώνονται σε τέσσερα ζητήματα που συνδέονται με ένα πιθανό πλαίσιο μετά το Safe Harbor. Πρώτα να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα είναι πιο ισχυρή και με πιο ισχυρή εποπτεία από την προηγούμενη οι ε, δεσμεύσει ε, χρηστή ε, διακυβέρνηση που έχει κάνει η Αμερικανική πλευρά θα πρέπει να τηρούνται και μάλιστα να είναι δεσμευτικέ. Δεύτερον, να διασφαλίσουμε ότι οι επιμέρους ε, παράπονα των Ευρωπαίων πολιτών θα τυχάνουν τους απαραίτητες επεξεργασίας. Και έτσι η συμμόρφωση και από τις αμερικανικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιούνται και να επιβάλλονται. Πώς, ε, τώρα το πώς θα πετύχουμε ακριβώς αυτή την κατάλληλη εποπτεία είναι ένα θέμα συζήτησης. Όμως κατά τη γνώμη μας η καλύτερη λύση θα ήταν να εμπλακούν αμέσως, άμεσα και ε, οι εθνικές αρχές ε, δεδομένων σε στενή συνεργασία και με τις αμερικανικές αρχές. Ε, χρειαζόμαστε όμως και σημαντικές ασφαλίσεις ότι η πρόσβαση στις δημόσιες αρχές περιορίζεται στα πλέον απαραίτητα και αναλογικά. Όπως γνωρίζετε και τα ανέφερε και προηγουμένως στο παρελθόν μάλλον η κυρία Γιούροβα, έχουμε δει σημαντικές ε, και πολλά υποσχόμενε εξελίξει το τελευταίο διάστημα για την Αμερικανική πλευρά. Πρέπει όμω να εξασφαλίσουμε ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι επαρκή. Ακόμα όμω διερευνούμε αυτή την κατάσταση. Τέλο, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι περιορισμοί στο νομικό πλαίσιο μεταφράζονται και σε πραγματικέ τροποποίησει ε, στα όσα σημαίνουν στην πράξη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό επαλήθευσης εκ των υστέρων που θα μας επιτρέπει να ελέγχουμε ότι ε, τυχόν διασφαλίσεις που θα λαμβάνουμε θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Χρειαζόμαστε λοιπόν περιοδική υποβολή εκθέσεων από τις Αμερικανικές επιχειρήσεις ε, για τον αριθμό των ετοιμάτων πρόσβαση δεδομένα επιτρέπεται και από το Freedom Act της Αμερικανικής Κυβέρνησης του 2015. Έχουμε ζητήσει από τους Αμερικανούς αυτή η υποβολή εκθέσεων να είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνία Safe Harbor. Θεωρούμε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν περισσότερες εκθέσεις ειδικά για το Safe Harbor από τις Αμερικανικές Αρχές. Στη Washington έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος για να ξεκαθαρίσουμε καλύτερα τους περιορισμούς και τους μηχανισμούς εποπτείας σε φορά την πρόσφαση στα διαβασμένα αυτά δεδομένα και την χρήση αυτών των ε, δεδομένων από τις ε, δημόσιες αρχές για σκοπούς ε, δημοσίου συμφέροντος και εθνικής ασφάλειας. Ταυτόχρονα πρέπει να εργαστούμε περαιτέρω σε δύο κύρια ζητήματα. Διαφάνεια σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων για τα αιτήματα πρόσβαση στα δεδομένα και ε, ο μηχανισμός σε ό,τι αφορά τις αυτοπιστοποιούμενες ε, επιχειρήσεις. Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση και στην Γερουσία και στο Κογκρέσο για να ε, υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και υπάρχει όθηση και δυναμική και από τις επιχειρήσεις. Γιατί και εκείνη η πλευρά θεωρεί πολύ σημαντικό στοιχείο και για την προώθηση της ιδιωτικής σφαίρας ζωής και στις ΕΠΑ. Ταυτόχρονα δεν είναι πάντα εύκολες οι συζητήσεις αυτές, οι συνομιλίες. Και πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μία σειρά λύσεων για να έχουμε ένα εύρο στο πλαίσιο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε επιτυχία να ολοκληρώσουμε τις συνομιλίες στις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, Βάσει και τη δικαστική απόφαση, ποια η Αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη κατανόηση και ε, με δημιουργικό και φάνταστο τρόπο να βρούμε νέες ε, λύσεις ε, στο στενό αυτό χρονικό πλαίσιο που έχουμε στη διάθεσή μας. Βέβαια είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Βεβαίω, ε, τη στιγμή που η Επίτροπο Γιούροβα βρισκόταν στη Ουάσιγκτον, είχαμε και τι ε, τραγικέ επιθέσει στο Παρίσι, που αποτελούν μεγάλη πρόκληση για μα και πολλά κράτη-μέλη θέλουν να ενισχύσουν, να ενδυναμώσουν του κανόνε ασφαλεία του. Ε, θέλουν ενισχυμένη συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση τη δημοκρατία. Αυτό καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η εξισορρόπηση της προστασία δεδομένων με τα συμφέροντα εθνική ασφαλεία. Όμω, επιβεβαιώνει και την αναγκαιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ να συνεργάζονται και να άρουν τυχόν προσκόμματα ε, σε αυτή τη διαδικασία. Κλείνοντα, να πω ότι μόνο ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο με συγκεκριμένε δεσμεύσει και δυνατότητε εφαρμογή τους ε, μπορεί να διασφαλίσει στην πράξη ε, αυτό το επίπεδο προστασία δεδομένων που επιθυμούμε και το οποίο ε, ορίζεται και από το, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί προστασία δεδομένων. Αυτό χρειαζόμαστε και επί αυτού εργαζόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μωρίγιο. Είναι πολύ σημαντικά τα όσα συμβαίνουν για το Safe Harbor, αγαπητοί συνάδελφοι, και είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσά θέλουν να λάβουν το λόγο τώρα. Θα ξεκινήσω με τον σκιώδη συγκητή για τη δέσμη μέτρων για την προστασία δεδομένων και από εκεί και πέρα θα ε, μιλήσουν οι υπόλοιποι συντονιστέ και μετά τα, οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ο κύριος Βος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εσάς κύριε Μόριο για τις εξηγήσεις που μας δώσατε για τα όσα συμβαίνουν και τις επιπτώσεις των όσων προγραμματίζεται. Όλα αυτά ακούγονται καλά. Δεν υπάρχει και διερμηνία, λέει ο μελητής. if Yeah. Nochmals vielen θα ήθελα εκ νέου να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας. Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ καλά και συνεκτικά και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι έχετε τόσο ευρία ε, παρουσίαση σε ό,τι αφορά το θέμα της μεταφοράς δεδομένων σε τρίτες χώρες. Θεωρούμε ότι αποτελεί ένα ουσιαστικό και κεντρικό θέμα και στο μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω καταρχάς πόσο πιθανό είναι πραγματικά μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου να πετύχουμε όντως κάτι και πώς σκοπεύετε να πετύχετε την αρμόνιση στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να την εγγυηθείτε. Άλλωστε υπάρχει δυνατότητα μέσω των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων να υπάρξει μία ερμηνεία. Θα θέλαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε με τον κανονισμό εναρμονισμένο δίκαιο, στη συνέχεια το FTC. αποτελεί μια ευκαιρία να ρέχουμε με πιο αυστηρό τρόπο και να διδραματίσουμε ένα πιο κεντρικό ρόλο. Και τέλος, έχετε την αίσθηση ότι στις ΕΙΠΑ υπάρχει κατανόηση του πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και το πόσο γρήγορα πρέπει να προχωρήσουμε όπως και εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Η κυρία Λάρσεν από πλευρά Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ και για αυτή την παρουσίαση. Όπως ε, γνωρίζετε, φτάνουμε πλέον στο τελευταίο στάδιο για το νέο κανονισμό για την προστασία δεδομένων και έχει ήδη συμπεριληφθεί σε αυτόν στο μέτρο του δυνατούν και η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση και τα όσα προβλέπει. Η ερώτηση μου είναι εξής επειδή έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά και αν κατάλαβα καλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά για να καταλάβει όλες τις συνέπειες αυτής της δικαστικής απόφασης. Τι μπορείτε να μας πείτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κατάλαβα καλά, ε, μετέβει η κυρία Γιούροβα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ελπίζω να μας αναφέρει και τι έχει γίνει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πόσο σοβαρά λαμβάνουν υπόψη τους αυτή την απόφαση. Διότι η δικαστική απόφαση αποδεικνύει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κατάλληλο επίπεδο προστασίας ε, στι Ηνωμένε Πολιτείε. Μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα λοιπόν από αυτού. Τι διάθεση υπάρχει και τι περαιτέρω ε, κινήσει σκοπεύει να κάνει η Αμερικανική πλευρά η Σόφη Ινεντβέλ που είναι σκιώδης των φιλελευθέρων για το μέτρων για την προστασία δεδομένων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η συνάδελφος προηγουμένως, διότι αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Τι προτίθεται να κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε προ το συμφέρον του, όχι γιατί του ζητούμε εμεί, αλλά γιατί θέλουν να συνεργαστούν με την Ευρώπη. Ε, δεν θα πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Υπάρχουν κάποια ζητήματα κατά την άποψή μου με όλο το συμβασμό και την εκτίμηση που σας έχω κύριε Φωνσέκα Μωρίγιο ε, και ε, τα όσα κάνει και η κυρία Γιούροβα. Αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο συνόδη κορυφή. Γιατί θεωρείται ένα διοικητικό θέμα. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό το οποίο συζητούμε είναι το γεγονός ότι πρέπει οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους. Αυτό λέει στην ουσία ο δικαστής. Άσχετο με το τι νιώθετε για την πολιτική σκοπιά, αυτό πλέον αποτελεί νομολογία. Τελεία και παύλα. Προκειμένου λοιπόν να συνεργαστούμε μαζί μας, θα πρέπει να υπάρχει ένα ε, νομικό πλαίσιο που να τους το επιτρέπει. Δεν κάνουμε ε, με όποιον να είναι απλώς και μόνο γιατί είναι καλοί φίλοι μας άκουσα αυτά που είχατε να μας πείτε και όντως μπορεί να είναι και όλα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά δεν αναφέρονται καθόλου στην ουσία. Ασχολούμαστε μόνο με τα παρελκόμενα. πρέπει να γίνεται περισσότερα παλίδες να έχουμε περισσότερες εκθέσεις, αλλά δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Δεν μας είπε ο δικαστής ότι δεν είχαμε αρκετές εκθέσεις ε, για τον αριθμό των ετοιμάτων πρόσβασης. Ο δικαστή είπε απλώ ότι τα δεδομένα μα δεν είναι ασφαλή στι Ηνωμένες Πολιτείες γιατί οι Αμερικανικέ Υπηρεσίε πληροφοριών έχουν απεριόριστη πρόσβαση. Αυτή είναι η ουσία τη απόφαση του δικαστηρίου. Τι κάνουμε λοιπόν εμεί εμεί εδώ, τι συζητούμε, δεν είναι σοβαρή η στάση μας. Ποια θα είναι η πραγματική λύση, θα υπάρξει κάποια λύση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι διατεθειμένες να μετακινηθούν, γιατί αν δεν είναι διατεθειμένες να μετακινηθούν, έχει καλώς ε, επιλογή τους, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την ε, διαβίβαση δεδομένων. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι η προστασία των δεδομένων είναι ε, το αγαπημένο παιχνιδάκι κάποιων ε, αριστερών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι όμως έτσι. Πρόκειται για δικαστική απόφαση και αναφέρεται στο δικαίωμα για τη ζωή, την ελευθερία έκφρασης και την καταδίκη ε, των βασανισμών. Είναι θεμελιώδης δικαίωμα. Δεν μπορεί απλώς κάποιος να το κάνει μια διαπραγμάτευση γιατί ε, μας βολεύει και νομίζω Εάν ε, είχε γίνει κάτι αντίστοιχο για την απαγόρευση του βασανισμού, θα το αντιμετώπιζε με τον ίδιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρόκειται για συμφωνία με τι ΗΠΑ, πρόκειται για μονομαρή απόφαση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε μα παρέχουν ή όχι κατάλληλο επίπεδο προστασία. Ο δικαστή λέει όχι. Επομένω, τι δυνατότητες πίεσης έχει η Ευρωπαϊκή επομενω τι δυνατότητε πίεση εχει η ευρωπαικη επιτροπη να πείσει τι ΗΠΑ ότι αν θέλουν να κάνουν δουλειέ με την Ευρώπη θα πρέπει να παρέχουν αντίστοιχο επίπεδο προστασία δεδομένων. Αυτή είναι η ουσία. Ούτε εκθέσει, ούτε αποζημιώσει, ούτε δεσμευτικά μέτρα, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η ουσία. Ωραία, ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόνι τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή. Νομίζω ότι όλοι κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί μια λύση μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, αλλά αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω για τρεις λόγους. Καταρχάς, οι προσδοκίες, οι δικές μας και της ομάδας του άρθρου 29 για να ολοκληρωθούν οι προσωρινές ε, λύσεις τέλη του Ιανουαρίου Κατά δεύτερον, δεν έχουμε ιδέα για το πώς μπορούμε να πιέσουμε τους συναδελφούς από τις είπα, όχι μόνο να μιλάνε, αλλά να παρουσιάσουν πραγματικές λύσεις μέχρι τέλη Γενάρη. Και τρίτο θέμα που έχει να κάνει και με τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερως για τις μικρές επιχειρήσεις, για τις οποίες είναι πολύ δύσκολο να σέβονται όλους αυτούς τους όρους που προκύπτουν από τις ρήτρες. Άρα, από τη μία έχουμε το αισιόδοξο σενάριο, από την άλλη τι πρέπει να κάνουμε. Τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη του Γενάρη και μετά, όταν θα υπάρχει πραγματικά λύση. Και θα είναι έντονη η πίεση και από τη ΣΥΠΑ και από την ομάδα άρθρο 29. Ευχαριστώ. Η κυρία Σίπελ τώρα, η Μπρικίτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ προσεκτικά άκουσα πόσα έχουμε ακόμα να κάνουμε, πόσο υψηλές είναι οι προδιαγραφές της δικαστικής απόφασης ΣΡΕΜΣ, πόσα πολλά έχουν να τελευκανθούν και παράλληλα ακούω φήμες ότι για να είμαστε έτοιμοι τα τέλη Ιανουαρίου πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες τέλη Δεκεμβρίου. Αυτό με εκπλήσει. Τι θέλουν να κάνουν λοιπόν οι ΙΠΑ με την Ευρώπη. Αν μιλάμε για το safe harbor, για τον ασφαλή λιμένα, μιλάμε για επεξεργασία των δικών μας δεδομένων. Να είμαστε σαφείς. Οι επιχειρήσεις συλλέγουν δεδομένα άκρητα και χωρίς έλεγχο για το άτομο μου για παράδειγμα και μετά κάνουν ερμηνεία των δεδομένων αυτών. Η ερμηνεία των δεδομένων αυτών έχει ήδη συγκεκριμένες επιπτώσεις για τα άτομα και όχι μόνο μαζική, μαζικός βομβαρδισμός με διαφημίσεις τις οποίες δεν με επιθυμούν, αλλά το γεγονός για παράδειγμα ότι δεν παίρνουν δουλειές, δεν παίρνουν δάνεια, δεν μπορούν να πετάξουν οι άνθρωποι αυτοί ή ενδεχομένως να έχουν αρνητικούς όρους για τη χορήγηση των δανείων τους. Το θέμα των προσφυγών είναι πάρα πολύ ευαίσθητο γιατί στην ουσία δεν έχει ε, κοινοποιηθεί ο λόγος για τον οποίο υπόκειται το άτομο αυτό τις αρνητικές συνέπειες. Δεν μπορεί να γίνει λοιπόν ανάλυση του επίπεδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Πώς θα ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ανάλυση και πώς είναι δυνατόν να έχει ολοκληρωθεί τόσο σύντομα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των δεδομένων στη ΣΥΠΑ. Εγώ αναρωτιέμαι, μας φτάνει Μα φτάνει το γεγονός ότι η ΕΠΑ ή κάποια μεμονωμένη αρχή, υπηρεσία, επιχείρηση μας αναφέρουν το τι κάνουν. Αυτό γινόταν και στην παλιά συμφωνία Safe Harbor. Το θέμα όμως είναι, μπορούμε να τους εμπιστευτούμε, μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτές τις εκθέσεις για την τήρηση των προδιαγραφών για την προστασία των δεδομένων. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζονται πιο πολλές ε, διασφαλίσεις και σήμερα θα ήθελα πιο πολλές πληροφορίες. Περίμενα πιο πολλές πληροφορίες για το πώς διεξαγάγεται ο έλεγχος αυτός και η συνεργασία αυτή. Ευχαριστούμε, Μπρικίτ. Ο κύριος Λόκος Αγγιλάρ. Συμφωνώ με τα μηνύματα ανησυχία που ανέφεραν οι προλαλήσαντε, αλλά θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπηρεσίε του υπολόγισαν ποιε είναι οι συνέπειε αυτή τη ε, απόφαση του δικαστηρίου και σε άλλα ζητήματα που είναι ευαίσθητα. και μάλιστα έχουν ως κεντρικό θέμα την αποδυνάμωση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως είναι εγγεγραμμένα στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συνήθως οι δικαστικές αποφάσεις έχουν και ένα δογματικό περιεχόμενο το οποίο υπερβαίνει την ίδια την υπόθεση και ε, υπερβαίνει και τη συγκεκριμένη την υπόθεση επί της οποίας αποφάνθηκε. Και σε αυτή την περίπτωση λέγεται ότι είναι ασύμβατο με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο διότι αποδυναμώνει τα ε, δικαιώματα τα οποία περιλαμβάνονται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση λοιπόν του Συμβουλίου που σχετίζεται με τον μηχανισμό διαβίβασης δεδομένων αυτό το οποίο αποκαλούμε safe harbor ε, στο Ηνωμένο, στις Ηνωμένες είναι το περιεχόμενο της ε, απόφασης. Αλλά αυτά συνήθως προβάλλονται και σε άλλα ευαίσθητα ζητήματα. Και εκεί έχουμε αντίστοιχα αποδυνάμωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα του άρθρου 8 ε, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Υπάρχουν κάποιε υποθέσει οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστέ στην κοινή γνώμη και δεν έχει υπάρξει κάποια προληπτική συζήτηση σε βαθμό που κανείς ακόμα δεν γνωρίζει ποιο είναι το αρμόδιο δικαστικό όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσε να ε, συζητήσει το προδικαστικό ερώτημα το οποίο έχει καταλήξει τελικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Συνήθως όμως αυτές οι αποφάσεις έχουν και συστημικές επιπτώσεις σε αντίστοιχες συμφωνίες διαβίβασης δεδομένων σε τρίτες χώρες, οι οποίες εφαρμόζοντας την ίδια νομική λογική θα κριθούν άκυρες. Ο είτε πρόκειται για απόφαση του Συμβουλίου είτε για οποιοδήποτε άλλο νομικό μέσο. Θα ήθελα λοιπόν να μας ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συνέπειες υπάρχουν και ποιες είναι οι συστημικές επιπτώσεις της απόφασης όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτικότητα των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ, Χουαν Φερνάντο. Η Άννα στη συνέχεια σε ένα σεμινάριο που είχε διοργανωθεί στο πλαίσιο μια αντιπροσωπεία ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είπα πριν από πολλά χρόνια ακριβώ για την προστασία δεδομένων, κατάλαβα ότι δεν υπάρχει απολύτω καμία προστασία δεδομένων ε, στι ΗΠΑ. Και δεν είναι μόνο το θέμα της ε, NSA, γιατί εκεί υπάρχουν και ζητήματα ασφάλειας, αλλά είναι ευρύτερο. Οποιοςδήποτε στις ΗΠΑ μπορεί να φτιάξει μια βάση δεδομένων με τα δεδομένα που έχει διάθεσή του και μετά να την πουλήσει. Και μάλιστα Μα ενημέρωσε, υπήρξε δηλαδή παρουσίαση και από έναν ε, προηγούμενο πρώην υπάλληλο του Κογκρέσου που γνώριζε ακριβώ αυτά τα ζητήματα. Πώ μπορεί κάποιο να φτιάξει μια τέτοια βάση δεδομένων και μετά να την μεταπολίσει. Τελικά δηλαδή δεν μαθαίνουμε τίποτα από όλη αυτή την υπόθεση. Τώρα, υπό το φως και της νέας δικαστικής απόφασης, τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ήταν απόφαση της Κομισιόν που βρέθηκε στη βάση ακριβώς ε, της ε, συμφωνίας Safe Harbor το 2000. Ο κύριος Μωρίγιο, πότε κατάλαβα, είπε ότι πρόκειται ουσιαστικά για αρμοδιότητα των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων. Όμως, πολλά από τα κράτη-μέλη μας αδιαφορούν για τα όσα λένε και κάνουν οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να ξέρω, έχει έρθει σε επαφή με τις εθνικές αρχές αυτές για να διασφαλίσει ότι όντως υλοποιούν την δικαστική ε, αυτή απόφαση και στη χώρα μου, την Πορτογαλία. Εγώ ζήτησα από την Εθνική Αρχή να μου πει αν κάνει κάτι. Ναι, πράγματι μου είπαν ότι ενημερώνουν ότι υπάρχει αυτή η δικαστική απόφαση. Δεν απαγορεύουν σε καμία επιχείρηση ή μάλλον σε κανέναν να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Και ζήτησα έναν κατάλογο επιχειρήσεων, θυμόντουσαν έναν κατάλογο 125 επιχειρήσεων, κυρίως φαρμακευτικών, καλλιντικών κλινικών, ασφαλιστικών εταιριών, χρηματιστηριακών, Λουιβιτών Vuitton Πορτογαλίας, ζηδοποιείων, κινητών τηλεφώνων και το καθεξής. Όμως, αυτές ήταν μόνο επιχειρήσεις που είχαν αντοπιστεί μετά το 2010, όταν υπήρξε ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων. Δεν ξέρουν ποιες είναι οι υπόλοιπε επιχειρήσεις της προηγούμενης δεκαετίας. Και αυτά όλα στην Πορτογαλία που κατά τη γνώμη μου η Εθνική Αρχή Προστασία Δεδομένων κάνει ό,τι μπορεί. Όμω πραγματικά αμφιβάλλω κατά πόσο έχει αλλάξει κάτι πραγματικά στην πράξη. Βεβαίω, εντάξει, έχει υπάρξει προειδοποίηση, έχουν ειδοποιηθεί δηλαδή οι επιχειρήσει ό,τι αφορά τη δικαστική απόφαση. Αυτό όμω. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι, τι ακριβώ κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει όντω ότι οι εθνικέ αρχέ προστασία δεδομένων και οι κυβερνήσει τηρούν και σέβονται αυτή τη δικαστική απόφαση. Και συμφωνώ με τους αδέλφους που είπαν ότι αυτό θα πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα στις συνομιλίες μας με το Κογκρέσο. Γιατί προφανώς δεν πρόκειται να λυθεί αυτό αν το αφήσουμε μόνο στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Να υπενθυμίσω μόνο ότι Πολλά σημαίνουν στη λύπη βεβαίω, αλλά το χρονοδιάγραμμα που έχουμε είναι ιδιαίτερα φορτωμένο. 10 Ιανουαρίου έχει πει η κυρία Γιούροβα ότι θα επανέλθει. 10 Ιανουαρίου λοιπόν θα επιστρέψει και είπαμε ότι τότε θα πρέπει να μας απαντήσει και για τα όσα αναφέρουν ε, οι Αμερικανοί και τι γίνεται με τις ε, συνομιλίες. Όμως είναι ιδιαίτερα επίγον να έχουμε συμφωνία μέχρι τότε, μέχρι αυτή την προθεσμία. Γι' αυτό και υπάρχει αυτός ο προβληματισμός από τα μέλη κατά πόσο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τέτοια συμφωνία και τι θα γίνει μέχρι την καταληκτική αυτή ημερομηνία που είναι και πολύ σοβαρή. Α, Δεκέμβρη. 10 Δεκεμβρίου, συνέχεια λέω 10 Ιανουαρίου. Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου λοιπόν. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ λοιπόν να, αναλάβετε και να αντιμετωπίσετε αυτά τα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Πρέπει να ομολογήσω ότι ακούγοντας αυτά που μου είπατε αναρωτήθηκα Ποιε είναι οι πραγματικέ μας διαφορές όσον αφορά την ουσία αυτού του θέματος. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αρκετές από τις ερωτήσεις. Αλλά θα ξεκινήσω με την ερώτηση που αφορά το πολιτικό ή το διοικητικό επίπεδο που έθεσε η κυρία Ίνεντβελτ. Μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αμέσως Αμέσως όμως Η κυρία Μίχου, η προκάτοχός μου σε διοικητικό επίπεδο, η Επίτροπος Γιούροβα σε πολιτικό επίπεδο, αποφασίσαμε να διαμηνήσουμε στους Αμερικανούς ότι ε, έχουν αλλάξει τα πράγματα ε, εντελώς, ακριβώς λόγω της απόφασης. Γι' αυτό ακριβώς και η Επίτροπος ε, Γιούροβα με εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετέβη στη Washington πριν από 15 μέρες. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι δεν υπάρχει μια διοικητική τεχνοκρατική συζήτηση. Ε, το γνωρίζουμε απολύτως αυτό. Δεν πρόκειται για διαπραγμάτευση. Ε, διαπραγματευτήκαμε ε, δύο, για δύο χρόνια με τους Αμερικανούς, αλλά γνωρίζουν και συνειδητοποιούν πλέον ότι πρόκειται για πολιτικό ζήτημα και όπω είπε και ο Χωάν Φερνάντο Λόπεθ Αγγιλάρη, είναι ένα ζήτημα, α, είναι απλώς ε, θέμα κράτους δικαίου. Πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες μας για την προστασία των δεδομένων. Δεν ε, λέω ότι θα είστε ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι, αλλά απλώς σας λέω ότι συνοδητοποιούμε απόλυτα τι συνέπειες έχει το συγκεκριμένο ζήτημα. Ε, τώρα, θα προσπαθήσω να απαντήσω λίγο πιο συγκεκριμένα στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με το Ερώτημα του κυρίου Βοσ. Η ερώτησή σας λίγο πολύ ήταν αν έχουν συνειδητοποιήσει οι Αμερικανοί ότι μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Η απάντησή μου είναι ναι. Είναι πεπισμένοι ότι τα οικονομικά συμφέροντα που μας συνδέουν σημαίνει ότι πρέπει να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε επί νέας βάσεως ακριβώς λόγω των αλλαγών αυτών. Εάν τώρα ε, ξαναδώ το διοικητικό ζήτημα, οι συνάδελφοι που ήταν ε, στη Ουάσιγκτον, αν δεν κάνω λάθος, μου είπαν ότι οι, δυτικές, οι συζητήσεις είναι σκληρές μεν, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο το άνοιγμα που υπάρχει γιατί έχουν συνειδητοποιήσει το πολιτικό πρόβλημα. Θα ήθελα να είμαι λίγο σαφής. Η κυρία Γιούροβα στο θέμα αυτό θα είναι αδιάλακτη. Υπάρχει μια υποχρέωση και πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία πριν από το τέλος ε, Ιανουαρίου 2016. Η Επίτροπος Γιούροβα θα είναι εδώ σε 10 μέρες ε, για να σας ε, εξηγήσει τι πρόοδος υπάρχει. Μέχρι τώρα και τα τέλη Ιανουαρίου ε, είμαστε συνέχεια σε επαφή με τους Αμερικανούς για να συναντηθούμε είτε εδώ είτε στη Washington ή για παράδειγμα η επόμενη συνεδρίαση μάλλον θα γίνει στο Λονδίνο γιατί έτσι έχουμε καταφέρει να συνδυαστούμε η ΜΕΝ και η ΔΕ. Ε, υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα. Οι βασικές αρχές ε, είναι αυτές που σας εξήγησα στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Διαπραγματευόμαστε στην ουσία με τους Αμερικανούς πρέπει να είναι σαφές ότι μετά από την απόφαση της ΡΕΜΣ θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις οι οποίες θα είναι ε, υποχρεωτικές. Όσον αφορά το ερώτημα του κατά πόσον γίνεται σεβαστό το δικό μας σύστημα προστασίας των δεδομένων, εμείς διαπραγματευόμαστε με αντίστοιχη σκληρότητα, ε, επιτρέψτε με να πω, ε, κατά πόσον οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ευρώπη έχει δικαίωμα δικαστικής προσφυγής ε, και συζητούμε μαζί τους και τους λέμε ότι ανάγκη να απαντήσουμε στο θέμα της εθνικής ασφάλειας ε, είναι βάση των παραδόσεών μας, όπως είπε και ο κύριος Λόπος Αγγιλάρ, ε, με βάση και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι ανάλογες λοιπόν σε βασίες αυτών των αρχών και επομένω ζητούμε από τους Αμερικανούς να εφαρμόσουν αυτούς τους μηχανισμούς εκ των υστέρων. Δεν μπορώ να σας πω βέβαια με βεβαιότητα ότι θα βρούμε μια λύση σε κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα. Είμαι όμως πεπισμένο ότι το δικό μας το σημείο κίνησης, η προστασία των δεδομένων ως θεμελιώδες δικαίωμα, σημαίνει ότι πρέπει να συζητήσουμε ποιες είναι οι που πρέπει να υπάρχουν για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Σα είπα και προηγουμένω ότι χρειάζεται να συνεισφέρουν και οι δύο και συνειδητοποιούμε απόλυτα το συγκεκριμένο ε, γεγονός. Η κυρία Γιούροβα ε, θα επιδείξει πλήρη δαφάνεια, θα έρθει εδώ ε, και ενώπιόν σας είμαστε υπεύθυνοι όλοι και το γνωρίζετε. Ξέρετε ότι εμείς θα πρέπει να σας πούμε τι έχουμε διαπραγματευτεί. Νομίζω ο κύριος Βος και η κυρία Γκόμες αναφτά στο θέμα αυτό. Για το ρόλο των Εθνικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων υπάρχει οδηγία η οποία δίνει συγκεκριμένες αρμοδιότητε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Επιτροπή του άρθρου 29. Μετά την απόφαση REMS, συνεργαζόμαστε λοιπόν μαζί τους προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση και στη χειρότερη ε, ε, περίπτωση θα διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων. Και παρεπιπτόντος να σας πω ότι θα ήθελα να ξέρω και το λέει το εγγραφό για να ξέρω τι περιλαμβάνεται και ποιοι υπέγραψαν και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις. Δεν ξέρω, ελπίζω όμως ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία και να είστε βέβαιοι ότι η συμφωνία αυτή δεν θα είναι κατώτερη των προδιαγραφών μας. Κύριε Μπόνι, ε, μας είπατε ότι με αυτές τις διαπραγματεύσεις την απόφαση Σράιμς και ε, είναι πιο ισχυρή η κατάσταση. Θα υπάρχει πρόβλημα εάν δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι ουσιαστικό. Ξέρετε ότι δεν υπάρχουν ακόμα συγκεκριμένες απαντήσεις. Απλώς ε, το γεγονός ότι γνωρίζουμε όλα τα προβλήματα, διαπραγματευόμαστε με τους Αμερικανούς εδώ και δύο χρόνια και το μόνο που ζητάω είναι οι πολιτικές Αμερικανικές αρχές ε, να συνειδητοποιήσουν πλέον ότι έχει αλλάξει το παιχνίδι μετά από την απόφαση της το κατά πόσο θα επιστρέψουμε νικητέ, δεν το γνωρίζω. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά προκειμένου να τα καταφέρουμε και θα έχουμε χρόνο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου για να καταλήξουμε στις συμφωνίες. Ποιες είναι οι συνέπειες, κύριε Λόπεθε Γιλάρ, ποιες είναι οι συνέπειες σε σχέση με τις υπόλοιπε προτάσεις. Είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων συνεργαζόμαστε, εργαζόμαστε από αυτού, σίγουρα τα πάντα διακυβεύονται και συνειδητοποιούμε και τι συνέπειες μπορεί να έχουν τα συγκεκριμένα θέματα. Συνειδητοποιούμε όμως επίσης και ποιες είναι οι βασικές αρχές αυτής της διαπραγμάτευσης, χωρίς από την οποία, τις οποίες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και προσπαθούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά και πάλι χρειάζονται δύο πρέπει να ε, συνεχίσουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να τηρούμε την ίδια στάση ώστε να πείσουμε τους Αμερικανούς ότι το κοινό μας συμφέρον είναι να υπάρχει μια καλή συμφωνία safe harbor. Ε, δεν ξέρω αν είναι καλύτερο αυτό από την απόφαση που έχουμε. Δεν ξέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ενδεχομένω να επανέλθω στο θέμα αυτό, λέει ο Είναι πάρα πολύ σημαντικό άλλωστε και δυστυχώ θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη γιατί έχουμε ήδη μια καθυστέρηση. Έχουμε και τη συνάντηση στις 10 του μηνός, θα παρευρεθεί η Επίτροπος. Κατανοώ ότι πολλά ερωτήματα έχουν παραμείνει αναπάντητα. Συνάδελφοι, στις 10 του μηνός ε, θα τα θέσουμε αυτά τα ερωτήματα προς την Επίτροπο. Θα είμαστε και πιο κοντά στην προθεσμία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή για την παρουσίαση αυτή. And, ε, Ευχαριστούμε τον κύριο Μωρίλη και θα δούμε λοιπόν στι 10 του μηνό ε, και πάλι την Επιτροπή. Συνάδελφοι, λοιπόν, να περάσουμε πάρα αυτά στην ανταλλαγή απόψεων για, με την ε, Γενική Διεύθυνση Home. Να σα εξηγήσω από πού προήλθε το θέμα αυτό, ανταλλαγή απόψεων για την ευρωπαϊκή συνεργασία με την Τουρκία σε θέματα ασύλου, μετανάστευση και διαχείριση των εξωτερικών σύνορων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένη και της ε, συνάντηση των αρχηγών κρατών ε, της Κυριακής. Θέλαμε λοιπόν να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων για τις ε, συζητήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και των αποφάσεων που ελήφθησαν και πώς θα επηρεάσουν τα θέματα μετανάστευσης, ασύλου, ε, θεωρήσεων και το καθεξής τον Οκτώβριο πέρσι, μάλλον του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σε ό,τι αφορά την πρόοδο της Τουρκίας για την εφαρμογή του δικού χάρτη για την, ε, τις θεωρήσεις. Περιμένουμε και την έκθεση της Συνόδου του Ιουλίου και το ξέρω λοιπόν ότι οι συνάδελφοι γνωρίζουν και τι έγινε και την Κυριακή. 29 Νοεμβρίου σε ό,τι αφορά θέματα ασύλου και μετανάστευση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρούτη λοιπόν που βρίσκεται μαζί μας και έχετε το λόγο για να μας κάνετε την ενημέρωση και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Πολύ. Πρόεδρε. Υποτίθεται ότι θα ήμουν εδώ πιο νωρί ε, για να σας παρουσιάσω που βρισκόμαστε με την Τουρκία, αλλά κατά τύχη έρχομαι μετά τη σύνοδο. Καλή η χρονική συγκυρία λοιπόν. Θα προσπαθήσω, αν μου επιτρέπετε, να σας ε, παρουσιάσω το ευρύτερο πλαίσιο καταρχάς. Αυτό που πολλοί περιγράφουν ως ιστορική σύνοδο μεταξύ της Τουρκίας και των 28 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε με, το, με την Τουρκία και τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαντ, όλο ιδιαίτερος για να καταρτήσουμε ένα κοινό σχέδιο δράση σε ό,τι αφορά την διαχείριση της ε, μετανάστευσης. Αυτό ξεκίνησε λοιπόν στις αρχές Οκτωβρίου. Στόχο ήταν να συνεργαστούμε με την Τουρκία προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε καλύτερη διαχείριση των ε, ροών των μεταναστών, να δοθεί ένα τέρμα στην ε, παράνομη μετακίνηση μεταναστών και παράλληλα να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε πιο έντονα και πιο στεναρά με την Τουρκία για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών Όλα αυτά λοιπόν οδήγησαν στο κοινό σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία, όπω ονομάζεται, και το οποίο αποφασίστηκε με δημοψηφίσματα στις 15 Οκτωβρίου. Σε αυτό το κοινό σχέδιο δράσης λοιπόν ορίστηκαν μια σειρά από σημεία επί των οποίων πρόκειται να συνεργαστούμε με την Τουρκία. Και προφανώς υπήρχαν και αιτήματα από δικής μας πλευράς, υπήρξαν και αιτήματα από της τουρκικής πλευράς. Για να συνοψίσω, από πλευράς της τουρκικής κυβέρνησης υπήρχε αίτημα να υπάρχει να υπάρχει πολύ πιο τακτική συνάντηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Κατά δεύτερον, μια επιτάχυνση της ε, απελευθέρωσης ε, θεωρήσεων, κατά τρίτον ε, πρόοδος της διαπραγματεύσεις για την ένταξη και τέταρτον μεγαλύτερη χρηματοδότηση του έργου της Τουρκίας για την υποστήριξη των μεταναστών που έχουν καταφτάσει στην Τουρκία. Το σχέδιο δράσης λοιπόν αποφασίστηκε δημοψήφισμα στις 15 Οκτωβρίου. Μεταξύ 15 Οκτωβρίου και τη σημερινή ημερομηνία έχουν λάβει χώρα πολλές συναντήσεις με τις ε, τουρκικές αρχές για να δούμε πώς θα έπρεπε να εκτελεχτούν αυτές οι δράσεις. Και πλέον υπάρχει η αμοιβαία δέσμευση και από τις δύο πλευρές. Η χθεσινή σύνοδος μας επέτρεψε να συμφωνήσουμε για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, αλλά και για μια σειρά άλλων στοιχείων. Και Νομίζω ότι αυτό που είπαν πολλοί, ότι θα δοθεί νέα ενέργεια σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, αληθεύει. Ως εκ τούτου. Πλέον. Αναμένουμε από την Τουρκία να ενδυναμώσει την καταπολέμηση των παράνομων δικτύων διακίνησης ε, μεταναστών, να διασφαλίσει ότι θα είναι πιο λίγες οι παράνομες ε, αναχωρήσεις, να διασφαλίσει ότι οι διμερείς ε, όροι για την επιστροφή θα εφαρμοστούν καλύτερα και ότι θα λεφτούν ε, μία σειρά μέτρων για να επιτρέψουν την καλύτερη ένταξη των σύρων προσφύγων που βρίσκονται στην Τουρκία και που βρίσκονται υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας στην τουρκική οικονομία. Επίσης, ότι θα βελτιωθεί η εκπαίδευση των ε, παιδιών των οικογενειών από τη Συρία. Όπως σας είπα, υπήρξαν αιτήματα από τουρκικής πλευράς, ένα εκ των οποίων είναι η απέτηση δημιουργίας ε, ενός καταλήμματος για την ε, για τους πρόσφυγες. Επίσης, χθε ε, δόθηκε χρηματοδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα καταλήμματα προσφύγων. Αυτό δεν είναι για να πληρωθούν οι τουρκικές αρχές ε, για τη συνεργασία τους, το τονίζω, αλλά για να υποστηριχθεί να υποστηριχθούν οι δομές υποδοχή των προσφύγων στην Τουρκία. Κατά δεύτερον υπάρχει μια συμφωνία για την διεξαγωγή συνόδων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Τουρκίας με μια μορφή η οποία θα πρέπει να οριστεί κατά περίπτωση δις ανά και ότι οι σύνοδοι αυτοί θα συνοδεύονται από συνομιλίες σε υπουργικό επίπεδο πάντα βάσει του οδικού χάρτη και του σχεδίου δράση. Θα υπάρξουν και άλλε συναντήσει υψηλού επίπεδου, πολιτικός διάλογος, για να σας δώσω παραδείγματα. Κατά τρίτον, στα μέσα Δεκεμβρίου θα γίνει Υπουργική συνάντηση που θα ανοίξει το κεφάλαιο 17 υπάρχει δέσμευση να ανοίξουν και άλλα κεφάλαια στις διαπραγματεύσεις, αλλά σε πολλά από αυτά τα κεφάλαια πρέπει να πούμε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εντελεχής και εξαιρετική προκειμένου να εξεταστεί το κοινοτικό και εκτιμένο και να δούμε τι έχει αλλάξει από την τελευταία διαδικασία ελέγχου. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη λοιπόν η διαδικασία αυτή Τη εξέταση του κεκτημένου και της, ε, των σχετικών συζητήσεων. Αυτό λοιπόν περιλαμβάνει και το κεκτημένο ε, που αφορά την Επιτροπή σας, ε, κεφάλαιο 23 και 24, με σκοπό να ανοίξουν ενδεχομένως τα κεφάλαια αυτά την άνοιξη του 2016, αν και επιφυλάσσονται ακόμα τα κρατημέλη. Τέλος, αυτό φαντάζομαι αφορά και την Επιτροπή σας, καθώς και τον Επιτροπό Αβραμόπουλο και την Γενική Διεύθυνση Home, μια επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης του καθεστώτος ε, θεωρήσεων. Ήταν δύσκολες αυτές τι συζητήσεις, ξέρετε, γιατί σε μεγάλο βαθμό υπήρχε η αίσθηση ότι θα μπορούσε πολιτικός πώς να οριστεί μια ημερομηνία, αλλά παράλληλα έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε ότι για να κινηθούμε προς την απελευθέρωση από το καθεστώς θεωρήσεων έπρεπε να έχουμε πετύχει κάποια benchmarks. Έχουμε πάνω από 70 σημεία τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση από τις θεωρήσεις. Θα ολοκληρωθούν αυτά ενδεχομένως ε, γρήγορα τις επόμενες ημέρες και θα δούμε λοιπόν, γιατί ξέρουμε ότι πολλά νομοθετήματα είναι υπό κατάρτιση για, την, για τους ε, όρους αυτούς και περιμέναμε και την ανασυγκρότηση τη συγκρότηση σώμα του νέου κοινοβουλίου. Και πολλά στοιχεία θα πρέπει να εφαρμοστούν. Σκοπός είναι να κινηθούμε προς ένα καθεστώς ελεύθερο από θεωρήσεις μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους. Κάποιοι αναφέρουν τον Οκτώβριο του 2016 στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, αλλά σαφέστατα αυτό εξαρτάται από το πόσο θα μπορέσουμε να θεωρήσουμε ότι πληρώνται οι όροι προς την κατεύθυνση αυτή, τα benchmarks. θα πρέπει να καταθέσουμε πρόταση και θα πρέπει φυσικά να συμφωνήσουν και οι συνομοθέτες. Δεν υπάρχει φυσικά άλλη διαδικασία και άλλο περιθώριο. Τις τελευταίες εβδομάδες λοιπόν εργαστήκαμε σκληρά. Προκειμένου να τελεσφορήσουν οι συζήτησεις, οι συζήτησεις με την τουρκική πλευρά και για να διασφαλίσουμε ότι οι μεταναστευτικές ροές θα τυχάνουν χάνουν καλύτερες μεταχείρισης και διαχείρισης. Ξέρουμε ότι τις τελευταίες, τους μήνες είχαμε 600.000 αφήξεις μέσω των ελληνικών νησιών. Και ξέρουμε ότι όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις, μας απασχολούσαν πιο πολύ οι ροές από την Λιβύη προς την Ιταλία. Αυτό αποτελεί πλέον μόνο ένα κεφάλαιο από το πολλά κεφάλαια των μεταναστευτικών ροών. Αλλά πλέον υπάρχει μία σύγκληση απόψεων για την ε, κατανομή των ε, φορτίων αυτών. Έχουμε δύο εκατομμύρια στην Τουρκία Σύρους πρόσφυγες, 8 δις ε, δολάρια χρειάζονται από πλευρά της Τουρκίας για να ανταπεξέλθει στις συνεχείς αυτέ πιέσει. Και είναι σαφές ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι πρόσφυγες. Και υπάρχουν σαφείς αναφορές στα συμπεράσματα των ευρωπαϊκών και τουρκικών προγραμμάτων για την επανεγκατάσταση. Αυτό συνάδει και με τις γενικότερες συζητήσει που έχουμε. Και που σκοπό, σκοπό έχουν να προωθήσουν την νόμιμη μετανάστευση και όχι τη λάθρα μετανάστευση. Πρόεδρε, ελπίζω να μην μακρηγόρησα και ελπίζω να είναι και ζωηρή η συζήτηση που θα ακολουθήσει. Βεβαίω είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το ζήτημα και το χρονοδιάγραμμα. Όπω είπατε και εσεί, ε, η χρονική συγκυρία μάλλον ήταν εξαιρετική, γιατί είχαμε μόλι ε, την Κυριακή την Σύνοδο Όλα τα μέλη σχεδόν ε, που βρίσκονται εδώ έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ξεκινήσουμε με τους συντονιστές γιατί είχαν ζητήσει επισταμένω αυτή την συνάντηση, αυτή την ενημέρωση. Επομένω θα δώσω πρώτα στους συντονιστέ το λόγο και θα κρατήσουμε όσο γίνεται περισσότερο χρόνο για τα υπόλοιπα μέλη, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα. Αν μπορείτε να τηρήσετε τα δύο λεπτά, αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Σίπελ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Μετά αυτή την συνάντηση με την Τουρκία, εκκρεμούν ακόμα πολλά ζητήματα. Ακόμα δεν έχουμε και κάποιες συνεισφορές ορισμένων κρατών μελών για να χρηματοδοτήσουμε την υποτερμοστία για τους πρόσφυγες. Ε, λείπουν πόροι ε, προς το φρεγανικό καταπίστευμα, αλλά και από ό,τι φαίνεται το ζήτημα τη υπεράσπιση και προστασία των εξωτερικών ε, συνόρων προφανώς δεν απασχολεί όλα τα κρατημέλη εξίσου. Μπορείτε να μα πείτε από πού θα προκύψουν αυτά τα τρία δι. Δεύτερον, έχω κουραστεί να ακούω ότι η Τουρκία κάνει πολλά στον τομέα των προσφύγων. Αν συγκρίνεται ε, την οικονομική κατάσταση και την κατάσταση που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, νομίζω ότι ε, η κατάσταση στο Λίβανο είναι πολύ πιο βεβαρημένη. Πάντα όμως μιλούμε για την Τουρκία. Όταν λέτε ότι πρέπει τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν για καλύτερη στέγαση ε, και εκπαίδευση, πού θα γίνουν όλα αυτά, γιατί... Εγώ βλέπω ότι οι περισσότεροι από τους Σύρου πρόσφυγε δεν διαμένουν σε καταβλισμού, αλλά στις πόλεις της Τουρκίας. Πώς μπορούμε λοιπόν να οργανώσουμε ακριβώ τα πράγματα για να διασφαλίσουμε ότι θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα προ όφελο των προσφύγων. Μετά, οι Τούρκοι θα μπορούν ε, να ελέγχουν τα σύνορά του για να μην πηγαίνουν πλέον οι πρόσφυγε ε, στην Ευρώπη. Επίση, θα επιστραφούν ε, μετανάστε προ την Τουρκία, πάνω από 2 εκατομμύρια στην πορεία, αλλά δεν έχουμε ακούσει τίποτα για την επανεγκατάσταση. Τι συμβαίνει λοιπόν ως προς αυτό, είναι σημαντικό. Μέχρι τώρα, κανείς πρόσφυγας δεν έχει λάβει καθεστώς ασύλου στην Τουρκία. Είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή. Μετά, άκουσα ότι θα ανοίξουν κάποια κεφάλαια για την διαδικασία την ενταξιακή. Επί της αρχής ε, δεν έχουμε πρόβλημα. Το πολιτικό μου κόμμα πάντα έλεγε ότι θα πρέπει η Τουρκία να αποτελέσει τμήμα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ε, με τον Ερντογάν δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει τώρα και θα ήμουν ε, υπέρ του να πούμε πρώτα η Τουρκία θα πρέπει να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές και να ακυρώσει κάποιες τροποποίησεις που έκανε στο νομικό της πλαίσιο και μετά να ανοίξουμε τα νέα κεφάλαια. Γιατί η Τουρκία δεν είναι ε, ένα καλό πλαίσιο, μια καλή χώρα για τους Κούρδους, για τους νομικούς, για τους δημοσιογράφους και το καθεξής. Επομένως πρέπει να θέσουμε κάποιες προϋποθέσεις για να ξεκινήσουμε τα, τη συζήτηση για τα υπόλοιπα κεφάλαια. Και αυτό είναι κάτι που λείπει από εδώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να μην υπερβαίνετε τα δύο λεπτά. Η κυρία Στίβενς, παρακαλώ. Helga. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι σύντομη. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, η συστηματική ε, επαναπροώθηση μέσω pushback ε, προς την Τουρκία είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται. Ε, μετά αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν σε καταβλισμούς προσφύγων όπου θα μπορούν να ζητήσουν άσυλο. Στη συνέχεια υπάρχουν ε, θετικές ενδείξεις για τη μετακατάσταση στην Ευρώπη, ε, εφόσον δεν έχουν ακόμα επιβληθεί οι ποσοστώσεις. Αυτή ήταν και η πρόταση που είχε κάνει και η αντιπροσωπεία του ΕΝΒΕΑ. Και έτσι και αποφεύγουμε τους θανάτους στη θάλασσα και ο κάθε ε, πρόσφυγας έχει δικαίωμα να αιτηθεί άσυλο. Χθε συνήθι και εγκρίθηκε επισήμω και το σχέδιο δράση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Τρία δι λοιπόν για την ε, υποδοχή των ε, προσφύγων. Και έχουμε πλέον όλο το σχεδιασμό για την ολοποίηση του σχεδίου με στήριξη των υποδομών ε, και των pushbacks από την τουρκική ακτοφυλακή Όμως ε, δεν συμφωνούμε με την ε, απελευθέρωση των ε, θεωρήσεων, γιατί κάποιες φορές το τίμημα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Κυρία Σαζεντίνη, παρακαλώ. Α, είναι επί τη διαδικασία, Σεσίλια. Oh, I'm so... Α, συγγνώμη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως δεν κατάλαβα καλά τι είπατε, αλλά νόμιζα ότι θα έδινε το λόγο στου συντονιστέ πρώτα. Λοιπόν, πολλά υπόθηκαν ήδη από του ε, συναδέλφου και η Σίμπιλ ε, ρώτησε από πού προκύπτουν αυτά τα ποσά. Πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα. Κάποιοι θα έχουμε και έναν μακρύ κατάλογο ε, επιθυμιών, αλλά από πού θα προκύψουν από πού στο καλό θα έρθουν όλα αυτά τα χρήματα. Καλό θα ήταν να μα το απαντήσει αυτό κάποιο. Επίση, ισχύει αυτό που αναφέρεται στον τύπο ότι στι 14 και 15 το κεφάλαιο μόνο 17 θα ανοίξει η οικονομική και νομισματική πολιτική είναι ή όχι. Και σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση, ε, διαδικασία απελευθέρωση των θεωρήσεων μέχρι τα τέλη του 2016. Και πάλι μπορεί να το θεωρηθεί ως μία ευρύτερη επιθυμία, αλλά για την ε, προαγωγή της δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, η Τουρκία δεν τα πάει και τόσο καλά. Και όλοι επισημαίνουν πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει μία σε βάθος ε, δικαστική μεταρρύθμιση στην Τουρκία. Τι έχετε να πείτε επί τούτου, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και δεδομένου ότι ο Ερντογάν έχει ε, χειριστεί με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο τους πολιτικούς αντιπάλους προσφάτως. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αντιμετωπιστεί, λυθεί ή απλώς και πάλι τους ε, λαδώνουμε των εισαγωγικών για να το κάνουν ή πληρώνουμε για να καθαρίσουμε τη συνείδησή μας. Γιατί δείτε και στο λοιπόν τι συμβαίνει σήμερα. Όλοι οι πρόσφυγες είναι. Σε, σε αυτή την μικροσκοπική χώρα έχουμε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες. Επομένω, αν μιλούμε για τους πρόσφυγες, θα πρέπει να κάνουμε κάτι και στο Λίβανο που, είναι πολύ, που βρίσκεται σε πολύ πιο δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Έχει αντιμετωπιστεί αυτό, θα αντιμετωπιστεί στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σεσίλα. Ζητώ συγγνώμη δικό μου λάθος. Τώρα περνάμε στα μέλη με τη σειρά που ζήτησαν το λόγο. Η κυρία Μουσολίνη. Χωρίς ε, μικρόφωνο, κυρία Σαρτζεντίνη. Συγγνώμη, συγγνώμη, Τζούντιθ ε, Σαρτζεντίνη και μετά κυρία Βερζιά. Συγγνώμη, κυρία Βερζιά και μετά η Τζούντιθ Σαρτζεντίνη. Δεν είναι η μέρα μου σήμερα. Θα ήταν πολύ σοβαρό αν μιλήσει ε, πριν από μένα κυρία Σαρτζεντίνη. Εντάξει, τώρα δεν θα σκάσουμε, δεν είμαστε τόσο πολλάτρες. Θα ξεκινήσω την παρέμβασή μου λέγοντας ότι ε, και ε, εγώ ε, την ώρα που γινόταν η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας σκοτωνόταν ο Τεγκέρ Μπασίρ. Το Τεγκέρ Μπασίρ τον γνώρισα πριν από κάποια χρόνια. Ήταν ε, ακτιβιστής και πρέπει να μιλήσουμε και για αυτή τη δολοφονία και για τις επιθέσεις και τις δολοφονίες που γίνονται στην Τουρκία, ε, τις πρόσφατες επιθέσεις για παράδειγμα στην Άγκυρα. Η κατάσταση με την Τουρκία είναι περίπλοκη, υπάρχουν ε, ε αυστηρότερα μέτρα παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, περιορισμός της ελευθερίας έκφρασης, ε, ε, σχέσεις με το Ισλαμικό κράτος και τα κυκλώματα χρηματοδότησης που επιτρέπουν στο Ισλαμικό κράτος να έχει ίδιους πόρους χρηματοδότησης και αναρωτιέμαι ε, ε, για τον κύριο που μόλις ε, διόρισε Υπουργό Ενέργειας ο κύριος Ερδογάν. Υπάρχει κατά την άποψή μου κάτι πάρα πολύ περίεργο με αυτό το οποίο συμβαίνει με τι αφήξει των προσφύγων. Το είπαμε και το λέτε και εσεί σε κάθε περίπτωση ότι είχαμε επικεντρωθεί στι ροέ Λιβύη-Ιταλία. Και είπαμε ότι η εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχει κράτο στη Λιβύη. Αυτή τη στιγμή έχουμε τριπλάσιο αριθμό ανθρώπων που φτάνουν από την Τουρκία. Υπάρχει κράτο στην Τουρκία. Και επομένω τι συμβαίνει, γιατί αυτές οι χιλιάδες πρόσφυγες που έχουν τύχει τόσο καλή υποδοχή στην Τουρκία φτάνουν σοριδών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μένα αυτό είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό και πραγματικά εκπλήσωμαι που δεν ασχολούμαστε λίγο με το θέμα αυτό. Έχω εγώ κάποιες ιδέες ε, για το ποια είναι η σωστή απάντηση. Και μετά, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, η Human Rights Watch, ε, πιο συγκεκριμένα και η Διεθνής Αμνηστία, αναφέρθηκε σε πλήρη επαναπροώθηση από την Τουρκία στη Σύρων προς τη Συρία. Θα ήθελα λοιπόν να αναρωτηθούμε και γι' αυτό και για όλα τα καλά που υποτίθεται ότι έχει κάνει η Τουρκία ενώπιον των προσφύγων. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους που τηρείτε και το χρονοδιάγραμμα. Η Τζούντις ε, Σαρτζεντίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Μπίργκη Τσίπολ είπε πάρα πολλά από αυτά τα οποία ήθελα να πω. Με κάλυψε λοιπόν, δεν θα τα πω εγώ. Να συμπληρώσω, να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις εξαιρετικές εκθέσεις. Ενημερώνεται κάθε μέρα Ποιο κράτος μέλος πήλωσε για την υπατερμοστία, για το παγκόσμιο πρόγραμμα για τα τρόφιμα, για το καταπίστευμα για την Αφρική και ποιοι έχουν δεσμευτεί για επανεγκατάσταση ανθρώπων από την Ιταλία και την Ελλάδα. Τις απολαμβάνω, τις παρακολουθώ κάθε μέρα, αλλά αυτό δεν δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο σύστημα. Δημιουργεί εμπιστοσύνη στα δικά σας στατιστικά στοιχεία και όχι στο σύστημα. Εχθές υπήρχε μια συνάντηση με πρωθυπουργών, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για την Τουρκία και αναρωτιέμαι τι συμφωνία είναι αυτή. Ε, επανεγκατάσταση και θεώρηση διαβατηρίων ήταν θέματα τα οποία συζητήθηκαν εδώ πριν από χρόνια και υπήρχε και συμφωνία. Το Συμβούλιο όμως ήταν αυτό το οποίο δεν το προήθησε. Χρηματοδότηση 3 δις, πράγματι και εμείς θέλουμε να ξέρουμε από πού θα προέλθουν και τι ακριβώς θα γίνει και ε, σε τι θα τα δαπανίσουμε. Διότι έχουμε 2 εκατομμύρια πρόσφυγες και 3 δις ευρώ. Δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσό σε σχέση με το 1,8 παρεμπιπτόντων που δίνεται για την υπόλοιπη Αφρική μπορεί να θεωρηθεί ε, σωστό. Δεν υπάρχει κάποια ισορροπία, αλλά δεν είναι πολλά τα χρήματα. Φυσικά δεν ε, μιλάω στον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί εσεί εκπροσωπείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά νομίζω ότι πολλοί από εμά εδώ θεωρούμε ότι βλέπουμε μία συμφωνία πακέτο με την Τουρκία και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό ο οποίο επιφελείται. Αυτό όμω το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι σε καμία περίπτωση ωφελημένοι δεν θα είναι οι πρόσφυγε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κορά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από πέντε χρόνια, ένας κύριος ονόματι Καντάφη μας ζήτησε πέντε δις για να λύσει τα προβλήματα της μετανάστευσης από τη Λιβύη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απάντησε αρνητικά γιατί ο Καντάφη δεν ε, πληρούσε συγκεκριμένες ε, εγγυήσεις ε, για προστασία δικαιωμάτων αυτών των μεταναστών. Η πιο απλή ερώτηση λοιπόν την οποία θα ήθελα να θέσω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Τι εγγύησει για το σεβασμό των δικαιωμάτων μπορεί να μας δώσει ο Ερντογκάν όταν συστηματικά παραβιάζονται όλα τα πολιτικά δικαιώματα στην Τουρκία. Ε, αναφέρθηκε ο, ο Τούρκος, ο Κούρδος, συγγνώμη, δικηγόρος, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από δύο μέρες, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί από την αντιπολίτευση, οι ακτιβιστές ε, υπέρ των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οι οποίοι ε, δολοφονούνται ή την χάνουν επίθεση. Ε, τα τελευταία χρόνια δώσαμε δισεκατομμύρια κονδύλια προσχο, προενταξιακής βοήθειας στην Τουρκία για να προχωρήσει κάποια θέματα και εγώ έχω την εντύπωση ότι το θέμα τη προστασία των δικαιωμάτων στην Τουρκία δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Νομίζω μάλλον ότι είμαστε βέβαιοι ότι ο Ερντογάν είναι ένα πολύ καλό ε, ε, παίκτη στο διπλό παιχνίδι. Δεν μα δίνει καμία εγγύηση για αυτά τα οποία μα δίνει, παίρνει αυτά που θέλει και κατά πάσα πιθανότητα παίζει και σε διάφορα τραπέζια, κάποια εξ αυτών και επικίνδυνα. Επομένω, θα ήθελα να ξέρω τι εγγύησει έχουμε ότι αυτά τα τρία δι, τα οποία δεν είναι μεν πολλά, δεν επαρκούν κατά πάσα πιθανότητα σε σχέση με τις ροέ μεταναστών που έχουμε, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολλά χρήματα και δεν έχουμε κανένα ε, τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι θα δοθούν κατά Και ορισμένες φορές αφήνουμε τα πράγματα σε κάποιου ο οποίο δεν ενδιαφέρεται ε, για το πώς θα τα διαχειριστούν και τι θα τα κάνουν αυτά τα κονδύλια. Η κυρία Μουσολίνη στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ νόμιζα ότι σήμερα ερχόσασταν να μας πείτε ότι επιτέλους έχουμε αυτή τη συμφωνία. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία θα πρέπει να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρία δις, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει την απολευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων. Μα είναι δυνατόν. Εμείς δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη και τη, ε, όσα συνέβησαν. Μας το είπε λίγο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαίνεται σαν δεδομένη η συμφωνία. Είχαμε τη δολοφονία του δικηγόρου, την κατάρριψη του αεροσκάφου. Ε, και, αλλά το θέμα είναι ποιες είναι οι Εμείς θα δώσουμε χρήματα, ποιος θα κάνει έλεγχο. Έχουμε ανταλλαγή συνόρων ε, στην Τουρκία μεταξύ Συρίας, γίνεται ανταλλαγή όπλων, ανθρώπων. Εγώ είδα λοιπόν ανθρώπους, ε, δεν μπορώ να τους πω στρατιώτες, αυτούς που είχαν καταρρύψει το ρωσικό αεροσκάφος. Εγώ νόμιζα ότι ήταν τρομοκράτες και τελικά ήταν οι Τούρκοι. Πραγματικά εγώ ε, είμαι αντίθετη πάρα πολύ σε αυτή τη συμφωνία. Ο κύριος Δεπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να το πω αμέσω. Δεν εμπιστεύομαι και πολύ τον κύριο Ερντογκάν και διαφωνώ και με τις πολιτικές του ή λέει ότι είναι οι μόνοι που αντιστέκονται σε Ισλαμικό κράτος και αφήνει να περνούν από τα σύνορά τους αλεξέλεγκτα καύσιμα και όπλα, δεν κάνει τίποτα για τους πρόσφυγες. Έχω ένα μακρύ κατάλογο. Έχω το εξή όμως. Όσον αφορά τα τρία δι, διάβασα το επίσημο έγγραφο και λέει ότι κοστίζει 8 δι ε, στην Τουρκία ε, να ε, παρέχει πρόσφυγε. πρόσφυγες. Εδώ λέει 8 δις, είδα κάποιο άλλο έγγραφο το οποίο αναφερόταν σε 6 δι. Και πού είναι αυτές οι εκτιμήσεις βάσει των οποίων καταλήξαμε σε αυτό το ποσό. Και επίση, όπω είπε και οι συνάδελφοι, 500.000 ε, είναι στους καταλαβλισμούς που είναι λιγότερο και από αυτούς που είναι στη Λιβύη και στην Ιορδανία. Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτά τα τρία δις. Ε, τα, αυτά τα τρία δις πού θα δοθούν όμως, ε, τι δεσμεύσεις έχετε κάνει, για πόσα χρόνια για παράδειγμα. Δεύτερον, όσον αφορά την απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίων, εδώ πάλι έχω κάποια στοιχεία. Στην τελευταία έκθεση, και το είπατε κι εσείς, ε, υπήρχε πολύ μεγάλη ε, πρόοδος που έπρεπε ακόμα να γίνει σε 70 διαφορετικές κατευθύνσεις και θα απελευθερώσετε τις θεωρίες διαβατηρίων μέχρι ε, το τέλος του έτους. Επιτρέψτε μου ότι, να πω ότι με την κατάσταση που ισχύει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία ε, να σας πω το εξής. Δεν θα σταματήσουν τους πρόσφυγες, ε, ανέκδοτα σας λένε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ίσα ίσα ανοίγετε νέες πόρτες, θα αρχίσουν να έρχονται και από την Τουρκία. Ε, ελπίζω να συνειδητοποιείτε λοιπόν τι κάνετε. Τρίτον, η επαναπρόθεση. Η επαναπρόθεση είναι για ποιου, για τους Τούρκους που θα έρθουν σε εμά, για αυτούς οι οποίοι έρχονται παράνομα με εξαίρεση αυτών που έχουν καθεστώς πρόσφυγα. Ε, επίσης, υπάρχει μια άλλη πρόταση και εδώ εκφράζω μια προσωπική μου άποψη. Θα ήθελα να σας πω να ε, θεωρείται η Τουρκία χώρα καταγωγής. Στην Τουρκία για τους δημοσιογράφους, για τους νομικούς, για τους Κούρδους. Πριν μας πείσετε λοιπόν ότι θα μπορείτε να τη βάλετε στον κατάλογο των ασφαλών χωρών, θα πρέπει να κάνετε πολύ μεγάλες προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση έχω να κάνω για κάτι το οποίο για πρώτη φορά άκουσα μετά τη σύνοδο τη Κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε σε προηγούμενα συμβούλια. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη συνεργασία με την Τουρκία, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των ε, διακινητών και την καταπολέμηση των ε, οργανωμένων εγκληματιών. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλη κλίμακα αυτέ οι επιχειρήσει στο Αγίο Πέλαγο. Αναφέρθηκε λοιπόν αυτό, αλλά σε τι βαθμό και τι προβλέψεις, τι διατάξει ε, αποφασίστηκαν, σε τι βαθμό θα συνεργαστούμε με τι αστυνομικέ δυνάμεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τι έχουμε πετύχει έως ε, σήμερα στην καταπολέμηση των εγκληματικών αυτών ομάδων και τι μπορούμε να προσδοκούμε για το μέλλον. Θα ήθελα να ξέρουμε λοιπόν κατά πόσον προβλέπετε να διευρυνθούν αυτές οι επιχειρήσεις και πέρα από το Αγίο Πέλαγος, τον Εύξηνο Πόντο ενδεχομένω και σε ό,τι αφορά και την τρίτη περίοδο εφαρμογής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέιον. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με πολλού συναδέλφου. Ήθελα και εγώ να θέσω κάποια ζητήματα. Απλώ και εγώ θα ήθελα να φέρω και να αναφερθώ στι προποθέσει για να ανοίξουν ορισμένα κεφάλαια ό,τι αφορά την ανταξιακή διαδικασία, ιδίω ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όπω και συναδελφοί μου, και εγώ βλέπω ότι όχι μόνο δολοφονίε έχουν υπάρξει, αλλά και μάλιστα δύο δημοσιογράφοι έχουν φυλακιστεί. Κατηγορούνται για κατασκοπία και ο διευθυντή τη Κομεριέτ κύριε Γκιούλ. Επομένω, έχουν αλλάξει οι προποθέσει ε, για τα κεφάλαια στην αντεξή διαδικασία την τελευταία φορά που τα συζητήσαμε. Και ποια είναι η σύνδεση με την ετήσια έκθεση για την κατάσταση ότι αφορά την ανταξιακή διαδικασία που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο καιρό και δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή. Ο κύριος Τίμερμαν πήγε στην Τουρκία και εσείς κάποιες φορές ε, περιγράφεται μία απλή ζωή ενώ κάποιες φορές έχουμε πολύ διαφορετικές ε, απεικονίσεις ό,τι αφορά ιδίω ε, την εκπαίδευση και την υγεία ότι είναι δηλαδή πολύ άσχημες συνθήκες. Για τα τρία δι τα είπαν οι συνάδελφοι, θα το επαναλάβω και κάτι τελευταίο συμφωνώ με τόσο κύριο ο για το αντιστάθμισμα, ε, την, ε, τη συμπερίληψη της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των ασφαλών χωρών. Δεν αναφέρθηκε αυτό προηγουμένως και θέλω να το σχόλιο σας. Ευχαριστώ. Κυρία Σκάκιαλε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις μόνο σε ό,τι αφορά την επανεκατάσταση είναι απογοητευτικό το ότι δεν υπάρχουν αριθματικά στοιχεία ούτε οποιαδήποτε δέσμευση για τα μελλοντικά σχέδια επανεγκατάστασης. Ε. Αναφέρουμε και επαναλαμβάνουμε συνέχεια τις 20.000 ε, ανθρώπους για τα επόμενα χρόνια που θα επανεγκατασταθούν. Κάτι άλλο. Πείτε μας, ε, από τα εννέα κράτη-μέλη που παρέστησαν στην Σύνοδο με την Τουρκία, ποια ήταν αυτά τα, τα κράτη. Και ύστερα φαίνεται ότι υπάρχει μία σύγχυση για το κατά πόσον η Τουρκία θα θεωρηθεί ασφαλή χώρα ή ασφαλής τρίτη χώρα για το πώ θα επιστραφούν οι Σύριοι πρόσφυγες. Είναι ασφαλής χώρα προέλευσης η Τουρκία και ακούσαμε διάφορα και για τους ε, μετανάστε και για τι μειονότητες και κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ανακηρύξει την Τουρκία ασφαλή χώρα προέλευσης. Ευχαριστώ πολύ και την πύρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποιες ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου και μια παρατήρηση ίσως ως εισηγήτρια για την Τουρκία από πλευράς του Κοινοβουλίου. Τι το καινούριο υπάρχει σε ό,τι αφορά δηλαδή αυτή τη νέα πνοή που δίνεται στις διαδικασίες και στις διαπραγματεύσεις ε, ένταξη, ε, Πριν από ένα χρόνο, από ό,τι ξέρω, είχαμε βέτο για την έναρξη διαπραγμάτευσης του κεφάλαιο 17. Δεν ε, μειώσαμε τα κριτηριά μας. Τι ακριβώς καινούριο υπάρχει, πού έγκυται αυτή η πνοή. Γιατί εξ κατάλαβα, Ούτε η Γαλλία ούτε η Κύπρος χθες ήταν ε, το βέτο τους για την ε, διαπραγμάτευση των κεφαλαίων. Εμεί ήμασταν από πλευρά του Κοινοβουλίου πάντα ανοιχτοί στο άνοιγμα των κεφαλαίων. Στο κλείσιμο είμαστε πολύ αρνητικοί. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι θα πρέπει να πληρεί η Τουρκία όλου του όρου σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των παράνομων κυκλωμάτων λάθροδιακινητών. Όπω είπε και η Σκάι Κέλλερ, η Γερμανία θα ήθελα να γίνει και άλλη μια συνάντηση για την επαναγκατάσταση 4.000 ανθρώπων. Πείτε μας τι γίνεται. Σε ό,τι αφορά δε την επανεισδοχή και τη συμφωνία επανεισδοχή για τους υπηκόους τρίτων χωρών, υπάρχει συμφωνία είτε με την Τουρκία για τους Τύρκους υπηκόους. Αλλά αυτό θα αφορά και τους ετούντες άσυλο που περνούν από την Ελλάδα ή για παράδειγμα αν κάποιος περάσει από την Τουρκία στην Ολλανδία θα ισχύει και από αυτού του ατόμου η συμφωνία. Αν αφορά όμως μόνο την Ελλάδα, γιατί δεν επαρκεί η ήδη φυστάμενη διμερή συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Θα παρέχεστε λοιπόν στα ερωτήματα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ όλους του συναδέλφους για την συντομία τους και για τις ερωτήσει του. Ο κ. Βάλινχολτσερ τώρα. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι επί τη αρχή έχει νόημα να συνομιλούμε με την Τουρκία και πιστεύω ότι υπάρχει νόημα να υπάρχει και μια ρεαλιστική προσέγγιση στις συζητήσεις αυτές. Το αποτέλεσμα της Συνόδου όμως θεωρώ ότι είναι απογοητευτικό. Μεγάλες πομπόδεις ε, ανακοινώσεις, αλλά ουσιαστικά μικρό περιεχόμενο. Και υπάρχει το θέμα του περιεχομένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. και αυτό, η εκτέλεση του δικηγόρου αποτελεί κάτι το οποίο είναι αποτρόπαιο και δεν μπορούμε να το αποδώσουμε και στο ΠΚΚ. Παράνομες επιστροφές σύρων προσφύγων, Και παράλληλα η Τουρκία δεν επιτρέπει σε 170.000 Κούρτους να επιτρέψουν στα πάτρια του. τους. Αυτά δεν συζητιούνται βέβαια. Τουλάχιστον όχι στα συμπεράσματα. Αν συνεχίσουμε λοιπόν έτσι, θεωρώ ότι θα προκύψει και επιπρόσθετη ροή προσφύγων. Γιατί πολύ απλά πάρα πολλοί Κούρδοι δεν θα μπορέσουν να μείνουν στη χώρα τους. Και κάτι άλλο που δεν έχει να κάνει με την σύνοδο συγκεκριμένα, αλλά είναι σημαντικό για όλους μας. Το ακούσαμε ήδη. Γιατί δεν είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε εξίσου στα σοβαρά χώρες όπως ο Λίβανος, όπως και το Ιράκ. Γιατί η κατάσταση με τους πρόσφυγες είναι ακόμα πιο δραματική. Γιατί το συνομιλούμε λοιπόν με τις χώρες αυτές, προκειμένου να υπάρξει μια σταθεροποίηση της κατάστασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τόμας Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ συντομαρισμένα ερωτήματα. Πρώτον, ποιες είναι οι εγγυήσει που θα μας δώσει η Τουρκία για να διασφαλίσουμε ότι πράγματι αυτά τα χρήματα θα δαπανηθούν προς όφελος των προσφύγων και δεν θα τα χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να ενισχύσει τον προπολογισμό της σε ορισμένους τομείς. Η Τουρκία συστηματικά μας στέλνει πρόσφυγες ε, στην Ευρώπη. Έχω μιλήσει με πολλούς ε, γνώστες και είναι σαφές ότι είναι οργανωμένη αυτή η διαδικασία, προώθηση δηλαδή προσφύγων προς την Ελλάδα. Είναι μια χώρα που συνεχώς καταλύει τους δημοκρατικούς θεσμούς και μάλιστα εξέτασα και τις διατάξεις του ποινικού κώδικα σε ό,τι αφορά ε, την διακίνηση ε, μεταναστών και τις όλες διατάξεις που συνδέονται και με την ε, έκδοση ταυτοτήτων και το καθεξής και αυτό συνδέεται άμεσα και με την ε, ακριβώς την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Πρέπει να ασκήσουμε και εμείς πιέσεις, ούτως ώστε και η Τουρκία να αρχίσει ε, να τηρεί τις υποχρεώσεις σε ό,τι τις δημοκρατικές ελευθερίες. Και τέλο υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψει ένας ε, Τούρκος Κούρδο ε, Κούρδος ε, στην Τουρκία χωρί να έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη. Η κυρία Γκόμε, ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σα ρωτήσω γιατί δεν λειτουργεί το πρόγραμμα μεταγκατάσταση. Γιατί στην Πορτογαλία όλοι περιμένουν να έρθουν οι πρέσβειε, αλλά δεν έρχονται. Οι συνάδελφοί μου ανέφεραν τα πολύ σοβαρά ζητήματα που αφορούν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς όλα αυτά έχουν ε, παραλληλευθεί από το Συμβούλιο, ιδίω όταν έχουμε πολύ σημαντικά περιστατικά, όπως ήταν η δολοφονία του βουλευτή και νομικού, την φυλάκιση δημοσιογράφων και το καθεξής. Το ζήτημα της Κύπρου επίσης αμελείται. Ακούω ότι είναι στα σκαριά μια συμφωνία, αλλά θα έπρεπε να το συζητήσουμε περισσότερο. Μετά για την απελευθέρωση θεωρήσεων. Διάβασα μόλις ένα tweet που λέει ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί την προσφυγική κρίση για να πάρει μια συμφωνία υπέρ τη είναι ανήθικη, αλλά τουλάχιστον έξυπνη. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην άλλη, είναι και ανήθικη, αλλά και χαζή. Είπαν οι συνάδελφοι από πού θα προκύψουν τα τρία δις. Αλλά και πού θα πάνε, σας ρωτάω εγώ. Θα παρακολουθήσουμε την ε, πορεία που θα ακολουθήσουν ρωταω εγω θα παρακολουθησουμε την πορια που θα ακολουθησουν αυτα τα, κονδύλια. Σίγουρα όχι για να χρηματοδοτήσουμε τα τουρκικά νοσοκομεία που περιθάλπτουν ε, τζιχαντιστές ούτε για να χρηματοδοτήσουμε ε, τα οχήματα που μεταφέρουν το πετρέλαιο του ISIS ε, στην Τουρκία. Με τη συνενοχή της Τουρκίας. Σίγουρα όχι για να βοηθήσουμε την Τουρκία ε, να βομβαρδίσει τους Κούρδους. Γιατί να μην δώσουμε αυτά τα χρήματα σε σχολεία στο Ιράκ ή στο Λίβανο και γιατί να μεταδώσουμε για να ανοικοδομηθούν οι πόλεις που έχουν ανακτηθεί από τους Κούρδους και πραγματικά διακόπτουν ε, την γραμμή και αλυσίδα ε, του ISIS. Ευχαριστώ. Ε, Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ε. Κυρία Γκόμες, δεν ακούσαμε τίποτα για τη ρίζα, για τα αίτια που ο κόσμος φεύγει από τις χώρες τους. Αυτό αποτελεί ένα βασικό τμήμα του σχεδίου δράσης και μια βασική αιτία που ο κόσμος φεύγει από τις αιστείες τους, ο φόβος του Ισλαμικού κράτους. Και βλέπουμε λοιπόν ότι Τουρκία που υποτίθεται ότι καταπολεμάει τις αιτίες θα πρέπει να υποστηρίζει τους Κούρδους, όχι να τους ε, καταπολεμάει. Και θα ήθελα λοιπόν να ξέρω κατά πόσο συζητήθηκε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Κυρικός. Ευχαριστώ. Είναι πολύ δύσκολο κάποιε φορέ ε, να ζούμε με μια γείτονα χώρα όπω η Τουρκία, ιδίω όταν έχουμε αεροσκάφη τη που ε, παραβιάζουν νερό αεροχώρα μας κάθε εβδομάδα. Αλλά συμβιώνουμε και πραγματικά πιστεύουμε ότι η συνεργασία με την Τουρκία στο, στο θέμα τη προσφυγικής κλίση μπορεί να μα φέρει πιο κοντά στη λύση. Παρότι πολλέ φορέ κατακρίνουμε σφοδρά λοιπόν την Τουρκία, πιστεύουμε παρόλα αυτά ότι αυτή είναι η οδό που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Από αυτή τη θέση μέχρι να φτάσουμε στο άνοιγμα των επόμενων κεφαλαίων, για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Κατά τη γνώμη μου, το χειρότερο το οποίο θα προκύψει από αυτή την κατάσταση είναι ότι και πάλι Όσοι είναι υπέρμαχοι της Ευρώπης και θεωρούν ότι πράγματι η Τουρκία ανήκει στην Ευρώπη, η πίκοη της Τουρκίας, για άλλη μια φορά θα προδοθούν. Γιατί δεν λέμε ότι θα τα ξεπεράσουμε, θα τα λύσουμε όλα αυτά τα κεφάλαια, λέμε θα τα ανοίξουμε και θα ακολουθήσουμε τα κριτήρια. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να θεωρηθεί ότι πληρεί τα κριτήρια αυτών των κεφαλαίων. του δίνουμε ψευδεί ελπίδε. Αν θέλουμε να βρούμε κάτι να συζητήσουμε με την Τουρκία, ας εξετάσουμε το κάσους Μπέλη, το οποίο απειλεί να υπάρξει αν ε, εφαρμόσουμε το δίκαιο της θάλασσας και θα δούμε πότε θα είναι η Τουρκία έτοιμη για να ανοίξουμε αυτά τα κεφάλαια στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Δεύτερον, για να συμπληρώσω και το ερώτημα της ε, συναδέλφου Κάτι Πύρη. Ξέρετε ότι είχαμε 137.000 αιτήματα επιστροφών από την ελληνική κυβέρνηση προς την Τουρκία. Ξέρετε πόσοι μετανάστες έγιναν δεκτοί. ...3.833 από τις 137.000. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να μας δώσει οποιαδήποτε ελπίδα ότι θα είναι επιτυχής αυτή η συμφωνία για την οποία μας ενημερώνει τώρα η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Κύρκο. Δύο ακόμα ομιλητέ για να δώσουμε και λίγο χρόνο στον ε, ομιλητή να απαντήσει. Ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρου. Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ρούτε, νομίζω ότι και εσείς όπως και όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε να νιώσετε λίγο τι αίσθηση επικρατεί εδώ στην αίθουσα. Δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή να μιλήσουμε για ικανοποίηση, για διαφωνία ή ακόμα και την έκπληξη γιατί κάποιοι από εμά ε, ε, τελούμε υποσύγχυση για τον τρόπο με τον οποίο τόσο βεβαιασμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την ε, Τουρκία ανεξάρτητα από την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία. Θα έρθω στο προκείμενο. Περιμένουμε κάποιες συγκεκριμένε απαντήσεις. Υπάρχουν δύο εκφάνσεις αυτής της νέας κατάστασης που δεν είναι σαφείς. Καταρχάς, από πού προέρχονται τα χρήματα. Από πού θα προέλθουν αυτά τα τρία δις τα οποία θα διατεθούν στην Τουρκία και πώς θα είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτευχθεί ο στόχος ε, ε, για τον οποίο έχουν διατεθεί αυτά τα κονδύλια ο στόχος είναι να προστατεύσουμε τους πρόσφυγες από τη Συρία. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα δαπανηθούν νήλος ε, τα κονδύλια, όταν η ίδια η Τουρκία είναι πολύ σημαντικός παράγων στην περιοχή και φυσικά έχει και πολύ ε, μεγάλη αίσθηση εθνικής κυριαρχίας όπως ε, επέδειξε για τις προηγούμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γουίμπερκ τελευταία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για αυτές τις πληροφορίες ε, και θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς θα κάνουμε. Τρία δις ευρώ. Τα ακούσαμε επανειλημμένο σήμερα και 100 εκατομμύρια είχαμε μέχρι τώρα, 500.000 συγγνώμη είχαμε μέχρι τώρα. Ε, θα πείσουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν τα χρήματα, θα ε, αυξήσουμε τις ποσοστώσεις αυτή της λέσχης των λίγων πώς θα γίνει η κατανομή των κονδυλίων, θα υποχρεώσουμε ανθρώπους να μας δώσουν χρήματα, θα υποχρεώσουμε κράτη-μέλη υπό την απειλή κυρώσεων. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι οι Βρετανοί θέλουν να ανοίξουν τα μάτια των υπολείπων και να ε, μας δείξουν ότι υπάρχει λόγος που θέλουν να φύγουν. Ο κύριος Ρούτε, παρακαλώ πόσο χρόνο μου διαθέτετε, σας παρακαλώ κάντε ό,τι μπορείτε. Ξέρω ότι θέλετε να απαντήσετε σε ώρες ε, τις ερωτήσεις, αλλά έχουμε πάρα πολύ πίεση χρόνου. Θα προσπαθήσω, χωρίς να απαντήσω σε κάθε ερώτηση, να τις ομαδοποιήσω λίγο. Και αν παραλείψω κάτι, σας παρακαλώ υπενθυμίστε μου ή πέστε μου ακόμα και μετά ότι δεν σας απάντησα. Καταρχάς, χρήματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πρόταση για τη χρήση 500 εκατομμυρίων από ευρωπαϊκά κονδύλια και περιμένουμε και από τα κράτη-μέλη να διαθέσουν 2,5 δις ώστε να φτάσουμε στο σύνολο των 3 δισεκατομμυρίων. Από τα χθεσινά συμπεράσματα ε, υπάρχει σαφής δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά τα τρία δις, αλλά δεν ε, προβλέπεται από πού θα προέρχονται. Επομένως ε, υπάρχουν ακόμα κάποιες συζητήσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν για το θέμα αυτό. Υπάρχει όμως πλήρης δέσμευση όλων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων να εξευρεθούν αυτά τα τρία δις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ανέκαθεν έλεγε ότι μπορούμε να κινητοποιήσουμε κονδύλια από διάφορα ταμεία ε, περίπου 500 εκατομμυρίων. Δεύτερη ερώτηση που σχετίζεται με τα χρήματα. Ναι, είναι αποκλειστικά για τη χρήση ε, προς όφελος των προσφύγων. Κατά πάσα πιθανότητα θα προκύψουν από το καταπίστευμα το οποίο διαθέτουμε, το οποίο μας επιτρέπει να ε, βοηθήσουμε και πρόσφυγες από τη Συρία που πλήττονται και σε άλλες περιοχές ε, και δέχομαι αυτά που μας είπατε για τη Λιβύη και την Ιορδανία και φυσικά να σας πω ότι και αυτά τα θέματα συζητήθηκαν, όχι χθε με την Τουρκία, αλλά ε, τα γνωρίζουμε πολύ καλά και αυτά. Τώρα, το όλο θέμα της χρήσης των κονδυλίων θα το δείτε και με το καταπίστευμα για την Αφρική. Θα υπάρξουν συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Θα υπάρχει διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα τα εξετάσει και δεν είναι τρία δις που τα πετάμε έτσι στον αέρα. Δίνονται για πολύ συγκεκριμένα προγράμματα, για σχολεία, για κατασκευή υποδομών. Ε, δεν ε, μας ενδιαφέρουν μόνο οι καταβλισμοί αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε πόλεις. Ε, θα υπάρξει πολύ συγκεκριμένη παρακολούθηση λοιπόν των χρημάτων αυτών. Σα δίνω αυτέ τι απαντήσει. Δεν θα έπρεπε ω Γενικό Διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση HOME, γιατί είναι περισσότερο αρμοδιότητα άλλων συναδέλφων. Προσπαθώ λοιπόν να σα δώσω ό,τι έχω με βάση πληροφορίε που διαθέτω. Και με βάση την εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ μας. Για το θέμα των ε, νέων κεφαλαίων και το άνοιγμά τους. Αυτή είναι η περισσότερη ερώτηση που θα πρέπει να αποτανθεί στον ε, Επίτροπο Χάν ε, και σε άλλες γενικές διευθύνσεις. Αλλά επειδή εγώ ασχολήθηκα και με τις διαπραγματεύσεις διεύρυνσης 12 κρατών μελών, συμφωνώ απολύτως με την κυρία Πύρη ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το άνοιγμα των κεφαλαίων για να συζητήσουμε λήψεις στο σύστημα της υποψήφιας χώρας και εδώ συγκεκριμένα στην περίπτωση της Τουρκίας πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Εάν λοιπόν χρησιμοποιούμε τα κεφάλαια 23 και 24 στην πραγματικότητα θα τα χρησιμοποιήσουμε για να τους πούμε ότι αυτό δεν πάει καλά, αυτό δεν λειτουργεί, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ ε, κακή, ε, η εξαρτησία του δικαστικού σώματος είναι πολύ κακή και ούτω καθεξής. Ε, ε, το κλείσιμο του κεφαλαίου έρχεται όταν λέμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τις προϋποθέσεις. Ε, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ξέρω ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία τα τελευταία χρόνια από αυτού, αλλά η γενικότερη προσέγγιση είναι αυτή. Επομένως, καλό θα ήταν να ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση. Κάποιος, νομίζω, ήδη απάντησε σε κάποιον άλλον. Ε, ανέκαθεν υπήρχε πρόθεση να ανοίξει το κεφάλαιο 17, επομένως αυτό θα γίνει όντως στις 14 ή 15 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ε, στην ε, ε, διακυβερνητική διάσκεψη. Επανεισδοχή τώρα. Είναι σαφές ότι υπάρχει συμφωνία επανεισδοχής Ελλάδας-Τουρκίας Υπάρχουν και κάποιες διατάξεις επανειδοχής μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας. Υπάρχουν αντίστοιχες διατάξεις και μεταξύ Τουρκίας και Ρουμανίας. Κάποιες εξ αυτών είναι αποτελεσματικές, κάποιες άλλες όχι. Ε, να σας πω ότι αυτό είναι ένα από τα ουσιαστικά ζητήματα που συζήτησα και στην πρώτη Επιτροπή Επανειδοχής. Θα πρέπει να έρθω και να σας αναφέρω ε, τις εργασίες γιατί πρε, ε, μόλις συμφωνήθηκαν και τα πρακτικά της συγκεκριμένη συνεδρίασης και θα γίνει και μια δεύτερη συνεδρία της Επιτροπής Επανεισδοχής η οποία θα γίνει τον Ιανουάριο και θα θέσουμε αυτά τα θέματα επιτάπητος. Δεν θα ήθελα τώρα να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι σαφές ότι είναι προς το συμφέρον μας να διασφαλίσουμε ότι η Συμφωνία Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει και καλύπτει μόνο Τούρκους υπηκόους και θα πρέπει ταχύτατα να ισχύει και για υπηκόους τρίτων χωρών. Και αυτό ήταν και τμήμα των συζητήσεων ε, στα πλαίσια του σχεδίου δράσης ε, και της ε, επιτάχυνση της διαδικασία απελευθέρωση ε, θεωρήσεων διαβατηρίου και του σχετικού οδικού χάρτη. Να είμαστε λίγο σαφείς με την επανεισδοχή, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα άλλωστε. Δεν θέλουμε να στείλουμε πίσω ανθρώπους που έχουν κάνει αίτηση ασύλου. Θέλουμε να επιστρέψουμε ανθρώπους που δεν έχουν κανένα δικαίωμα να παραμείνουν ή που δεν έχουν πλέον δικαίωμα να παραμείνουν διότι οι διαδικασίες ασύλου έχουν περατωθεί και η απάντηση ήταν αρνητική. Και φυσικά αυτό θα ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη και όχι μόνο για την Ελλάδα. Επομένως, αυτό θα αφορά η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Τουρκίας για την επανεισδοχή και η συζητήση για την απελευθέρωση των θεωρώσεων διαβατηρίου θα γίνει για να δούμε κατά πόσον μπορούμε να έχουμε εφαρμογή της διάταξης για τους υπηκόους τρίτων χωρών αυτής της συμφωνίας και ανέκαθεν στο θέμα ε, της απελευθέρωσης των θεωρήσεων διαβατηρίων ως προϋπόθεση προκειμένου να μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε προς την απελευθέρωση των θεωρήσεων, ότι θα πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι λειτουργεί πλήρως η Συμφωνία Πανιζαχής και νομίζω ότι θα δείτε και σχετική διατύπωση και στα συμπεράσματα. Είναι λοιπόν αντιληπτό ότι η Τουρκία πρέπει πρώτα να εφαρμόσει τη διάταξη για τους υπηκόους τρίτων χωρών πριν μπορέσουμε καν να συζητήσουμε Προτάσει για απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίων, οι οποίε θα γίνουν σε, αυτό το στάδιο και χρειαζόμαστε και κάποια εμπειρία για την εφαρμογή πριν ε, μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ πιεστικό ε, για τη θεώρηση των διαβατηρίων. Δεν έχουμε απαρνηθεί τα 72 σημεία τα οποία εντοπίσαμε στην τελευταία έκθοση. Ε, είναι σαφές ότι πρέπει να εφαρμοστούν και συζητούμε και με την τουρκική πλευρά για το τι μπορεί να γίνει τώρα στην εφαρμογή, πόσο θα καθυστερήσει και υπάρχουν και πολλά ακαθόδη ζητήματα. Όπως γνωρίζετε υπάρχει το θέμα της προστασίας των δεδομένων Και επίσης, και αυτό περιλαμβάνεται στο κοινό πρόγραμμα δράσης, ε, θα ενισχύσουμε την αστυνομική συνεργασία για το λαθρεμπόριο και θα δούμε και πώς μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να υπάρχει και η προστασία δεδομένων και το κατάλληλο πλαίσιο. Αυτό είναι το ε, μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και κάτι από αυτού. Βλέπω λίγο τις ερωτήσεις σας. Η κυρία Κέλλερ ρώτησε για την επανεγκατάσταση. Όπως και εσείς και εγώ εφημερίδες διάβασα και χρειάζομαι κάποια περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχω είναι ότι μπορώ να περιοριστώ στα όσα λένε τα συμπεράσματα τα χθεσινά που αναφέρονται στα εθνικά προγράμματα επανεγκατάστασης και το υφιστάμενο πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει από εκεί και πέρα σε ποιο πλαίσιο θα γίνουν αυτά. Έχουμε ήδη ανακοινώσει ένα μόνιμο μηχανισμό επανεγκατάστασης ε, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπάρχει σχετική πρόταση, θα δούμε πώς θα ασχοληθούμε με αυτό. Αλλά νομίζω ότι μεσοπρόθεσμα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες προσπάθειες ε, για την επανεγκατάσταση από όσες κάνουμε αυτή τη στιγμή και θα έρθω με τα χαράς να σας πω που βρισκόμαστε. Επίσης ε, υπάρχει και συνεργασία σε εθνικό επίπεδο και μέσω της αρμοστίας βεβαίως ε, στις περιπτώσεις ε, που απαιτείται και αν δεν κάνω λάθος για το 2015 υπάρχουν δεσμεύσεις για 40.000 άτομα για επανεγκατάσταση. Δεν είμαι βέβαιος βέβαια για το κατά πόσον έχουμε ενημερώσει γι' αυτά. Ε, θα πρέπει να ρωτήσουμε και, ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το άσυλο την ΕΑΖΟ να δούμε αν μπορούμε να τα ε, προχωρήσουμε αυτά τα θέματα και να δούμε και τι δεσμεύσεις και τι εφαρμογή υπάρχει σε επίπεδο κρατών μελών. Είχαμε και πολλά άλλα γενικά ζητήματα που θίξατε, κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συνεργασία με την Τουρκία, είμαι βέβαιος και γνωρίζω ότι πολλά από αυτά είναι θέματα τα οποία συζητήθηκαν γενικότερα αλλά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και δεν θα ήθελα να επισέλθω εδώ σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές ότι πάντα έχουμε κατά νου την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα ήθελα εδώ να σας παραπέμψω στον οδικό χάρτη για την απελευθέρωση των διαβατηρίων των θεωρήσεων διαβατηρίων. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ορόσημα στο νοδικό αυτό χάρτη, ε, τα οποία θα βοηθήσουν και στη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Επίτροπό μου, τον κύριο Τίμπερμανς ε, και τον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά και για μας, ε, είναι ότι έχουμε σαφέστατα εμείνει στη δέσμευση να τηρηθούν τα ορόσημα του οδικού χάρτη για την απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων που θα βολτιώσουν και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιτόπου. Είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να επανέλθω βέβαια πολύ σύντομα για να συζητήσω και το θέμα των ασφαλών χωρών καταγωγής. Εξ όσων γνωρίζω δεν συζητήθηκε αυτό εχθές αλλά σίγουρα πρέπει να συζητήσουμε και ίσως με κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες ε, προσβλέπω σε αυτή τη συζήτηση κύριε Γκυγιόμ για το θέμα των ασφαλών χωρών καταγωγής. Πράγματι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία ξετάζουν και το άρθρο 38 και 39 τις οδηγίες για τις διαδικασίες ασύλου, για τις ασφαλείς τρίτες χώρες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι από αυτού και το κατά πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Αυτό το οποίο συζητάτε αυτή τη στιγμή είναι ο κατάλογος των ασφαλών χωρών καταγωγής που αφορά ανθρώπους που είναι υπήκοοι τρίτης χώρες, παραδείγματος χάρη Τούρκοι, και πάντα επιμένουμε ότι θα πρέπει να γίνεται εξέταση αναπερίπτωση. Είμαι βέβαιος όμως ότι αυτό θα το συζητήσουμε περισσότερο ε, σε κάποια άλλη στιγμή. Δεν είμαι βέβαιος ε, κατά πόσον κατάφερα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, προσπάθησα να αναφερθώ στα περισσότερα στοιχεία το οποίο αναφέρατε. Ζητώ συγγνώμη αν δεν απάντησα σε όλους σας έναν προς έναν. Ε, κατά πάσα πιθανότητα χρειαζόμουν δύο ώρες ε, για να το κάνω αυτό. Ε, ελπίζω να σας έδωσα κάποια στοιχεία. Ένα τελευταίο, κύριε Ρεπχέ. 8 δις δολάρια. Αναφέρονται σε 8 δις δολάρια και εμείς αναφερόμαστε σε ευρώ. Υπάρχουν κάποιες διαφορές λοιπόν για τα στοιχεία. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο, να τα δω όμω. Μπορούμε να τα εξετάσουμε και διμερώς. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ρούτα για τι απαντήσει που μας δώσατε. Ευχαριστώ και πάρα πολύ του συναδέλφου για τι ε, πολύ έστοχες ερωτήσει. Και ξέρω ότι θα χρειαστεί να επανέλθετε στα θέματα αυτά και είναι άλλωστε πάρα πολύ επίκαιρα και εκτιμούμε πάρα πολύ το χρόνο που μας αφιερώσατε. Um, Συνάδελφοι, βλέπετε ότι έχουμε καθυστερήσει. Συνάδελφοι, έχουμε καθυστερήσει, έχουμε και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία ενδεχομένως να μην τα προλάβουμε. 18 και 10 οι ψηφοφορίες. 6 και 10. Βρέξει χιονίσει θα γίνουν οι ψηφοφορίε. Να έχετε τι ηλεκτρονικέ σα κάρτε μαζί. Περνάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι το θέμα της, ε, για τους διαλόγους που θα μας ε, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα δικτύων. Και ο, ο κύριος Άλμπρεχτ είναι ο υπεύθυνο, θα πάρει το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή για την ενημέρωση για την οδηγία για τα δίκτυα και για τις πληροφορίες. Η αρμόδια καθήλυνα επιτροπή για το θέμα αυτό είναι η Επίτροπη ΕΜΚΟ. Ανδρέας Φάμπο, εισηγητής από το ΕΛΚ. Ο τριμερής διάλογος αυτός έχει λάβει χώρα κάποιες φορές ήδη. Έχουμε κάποια προβλήματα γιατί το Συμβούλιο σε κάποιες περιπτώσεις δεν παρουσιάζει τις πραγματικές του θέσεις και ως εκ τούτου έχουμε προβλήματα να ολοκληρώσουμε τον πρεμερή διάλογο αυτό παρά το γεγονός ότι πάντα προς την κατεύθυνση αυτή κινούμαστε. Πολύ σημαντική οδηγία που την έχει ήδη προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από κάποια χρόνια για την ασφάλεια IT και για τις ευαίσθητες υποδομές, τις ευάλωτες υποδομές. Βρισκόμαστε πλέον στην εξή ε, θέση. Ελπίζουμε να τελεσφορήσουν οι διαδικασίε και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει. 7 Δεκεμβρίου προσβλέπει ο εισηγητή ε, στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων από πλευρά του Κοινοβουλίου Είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τι διαπραγματεύσει από πλευρά του Συμβουλίου, όπω σα είπα, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα και σε κάποιε περιπτώσει πετυχαίνουμε μόνο μικρά βήματα και ενδεχομένω να χρειαστούν και άλλοι τριμερεί διάλογοι. Θα δούμε, θα δείξει, προσπαθούμε να πετύχουμε τη συμφωνία. Τι συμφωνήσαμε ω τώρα. Συμφωνήσαμε για το παιδί εφαρμογή ότι θα συμπεριλάβουμε πλέον και τις ψηφιακές υπηρεσίες, τους ψηφιακούς παρόχους, παρόχους διαδικτύου. Και εδώ όλοι διαπιστώνουμε Διαπιστώσαμε και πρόσφατα ότι υπάρχουν φυσικά ευάλωτες υποδομές. Το θέμα είναι πώς ε, θα οριστεί το πεδίο εφαρμογής, γιατί ουσιαστικά κάθε είδους τεχνολογία θα μπορούσε να παίξει το ρόλο της ε, σε ευάλωτες υποδομές, αλλά θα πρέπει να περιοριστούμε στις υποδομές και στους παρόχους που πραγματικά είναι ευάλωτες. Το Συμβούλιο είναι πολύ πιο περιοριστικό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τομείς που θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Αλλά στην τελική ανάλυση θα πρέπει να βρούμε μια λύση από πλευρά τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και ήδη, Πρόεδρε, ολοκληρώνω Στη γνωμοδότησή μα επικεντρωθήκαμε πάρα πολύ σε θέματα προστασία δεδομένων και καταφέραμε να προσεγγίσουμε. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, αλλά συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις κοινοποιήσεις, σε γέφυρες που θα πρέπει να υπάρξουν κοινοποιήσεις πάντα στις αρχές σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα. Αυτά λοιπόν ως τώρα και θα σας ενημερώσω αυτό το χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο έκτος τριμερής διάλογος προβλέπεται για τις 7 Δεκεμβρίου. Σε έκανα να βιαστείς λίγο γιατί έχεις να μας πεις και για το τι γίνεται για το επόμενο θέμα και εσύ και η κυρία Λόρες για το πακέτο προστασίας δεδομένων και τι γίνεται με τις τριμερείς ε, διαπραγματεύσεις. Να ακούσουμε πρώτα τον Γιάννη και μετά τη Μαριάννη. Ευχαριστώ πολύ Κλοντ. Πολύ σύντομα προσπαθούμε να κινηθούμε παρότι ξέρουμε ότι είναι τεράστιο το θέμα του κανονισμού προστασίας δεδομένων το οποίο μας έχει απασχολήσει εδώ και τέσσερα χρόνια περίπου, γιατί ξεκινήσαμε ένα ψήφισμα για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011. Από την... τον Ιανουάριο του 2012 υπέβαλε την πρόταση η Κομισιόν και εμείς υιοθετήσαμε σε πρώτη ανάγνωση πέρυσι την Άνοιξη και πλέον μπορούμε να ξεκινήσουμε τους τριμερείς διαλόγους. Ε, ήδη σας ενημέρωσα μια φορά μαζί και με την κυρία Λαρεστίν, Αμέσως μετά τις θερινές ε, διακοπές. Τώρα έχουμε ολοκληρώσει έναν γύρο διαπραγματεύσεων σχεδόν για όλα τα κεφάλαια. Τα μόνα που δεν έχουμε εξετάσει είναι οι τελικές διατάξει και οι διατάξει για τι εκτελεστικές και κατεξοδότητες πράξεις είναι τα τυπικά στο τέλος. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε όμως εξετάσει και όχι μόνο μία φορά. Σε ορισμένα ζητήματα τα έχουμε εξετάσει τρεις. Υπάρχει ένας κατάλογος εκρεμών ζητημάτων, όμως ε, είναι ήδη αρκετά περιορισμένος. Ακόμα εξετάζουμε θέματα που άπτονται της έρευνας, προστασίας δεδομένων στον τομέα της έρευνας, οι κύριε διαφορές είναι και πάλι ο ορισμός της έρευνας και οι δυνατότητες ε, που δίνονται για την επεξεργασία και πώς διαφέρουν από την προσέγγιση. Όμως δεν είναι ουσιώδες αυτές οι διαφορές. Θέλουμε να επιτρέψουμε την επεξεργασία δεδομένων σε αυτό το τομέα, αλλά βεβαίως όταν πρόκειται για ε, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως είναι η κατάσταση υγείας για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχουν ε, επιπλέον δικλείδες ασφαλείας όπως είχαμε πριν στο άρθρο 81 και τώρα ε, αναφέρεται στα, ε, στο άρθρο για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Επίσης, εξακολουθούμε να συζητούμε το πώς θα δίνεται η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων. Υπάρχει το ζήτημα της ρητής συγκατάθεσης και πότε αυτή είναι απαραίτητη, αλλά και γενικότερα σε ό,τι αφορά την ε, συγκατάθεση, πώς μπορεί να δίνεται και τη σύνδεση της συγκατάθεσης με όσα είναι απαραίτητα, αλλά και άλλες λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων. Και βεβαίως για να εξισορροπήσουμε τα πράγματα, έχουμε τις ε, δραστηριότητες επεξεργασίας ε, που έχουμε στον τομέα των συμβάσεων, αλλά και επανειλημμένης ε, χορήγησης της εγκατάθεσης, κάτι το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολο της αγοράς, αλλά συνδέεται και με τις ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, για παράδειγμα, που δραστηριοποιούνται στην ίδια ψηφιακή αγορά που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Τέλος, κάποιες διαφορές παραμένουν σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις ως προς την επεξεργασία δεδομένων για τους ε, υπεύθυνους επεξεργασίας και το καθεξής ιδίω ό,τι αφορά την ε, αρχή προστασία δεδομένων. μην επιμένουμε να, τουλάχιστον κάποιε από τι επιχειρήσει να διορίζουν έναν ε, αξιωματούχο, έναν υπάλληλο δηλαδή επεξεργαστή δεδομένων, όπω είναι υποχρεωτικό σε κάποια κρατημέλη. Το θεωρούμε σημαντικό και από πλευρά συναρμόνιση να έχουμε ενιαία πρότυπα σε όλη την αγορά. Ακόμα υπάρχει διαπραγμάτευση. Αλλά και για τις ε, κοινοποιήσεις γέφυρα, bridge notifications, μας έχουν πει ότι θα υπάρχει κάτι τέτοιο και για την προστασία δεδομένων, αλλά δεν είναι λυμένο κατά πόσο θα είναι απαραίτητο και αποχρεωτικό για κάθε περίπτωση ή αν θα υπάρχει μια ένδειξη επί του κινδύνου. Και μετά και το πρότυπο επιβολής κυρώσεων, που είναι και ένα από τα κύρια ζητήματα του κανονισμού. Θέλουμε εναρμονισμένη εφαρμογή σε όλα τα κρατημέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Έχουμε λοιπόν έναν μηχανισμό συνέπειας και συνοχής και έτσι θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους ε, οι αρχές προστασίας δεδομένων, αλλά υπάρχει και ο μηχανισμός κυρώσεων 2% ή 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης. Ε, είναι μια πρόταση που ακόμα εξετάζουμε σχεδόν για όλα τα υπόλοιπα θέματα πραγματικά μου φτάσει πολύ κοντά σε μια συμφωνία, πολύ πιθανόν στους δύο επόμενους γύρους πραγματεύσεων σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο να καταλήξουμε στη συμφωνία και για το πεδίο εφαρμογή ε, της ε, οδηγίας. Η κυρία Λονιστίν θα σας ενημερώσει τώρα για αυτά. Εγώ παραμένω αισιόδοξο Ελπίζουμε να έχουμε πολιτική συμφωνία και για τους δύο φακέλους του πακέτου πριν από τα τέλη της χρονιάς και προς υπενθύμησή σας είναι πολιτικός στόχος όχι μόνο του Κοινοβουλίου αλλά και της Επιτροπής και του Προέδρου της. Πρώτη και κύρια προτεραιότητα του σχεδίου εργασιών του ήταν ακριβώς να αριστικοποιηθεί αυτό το πακέτο μέσα στα τέλη του 2015 αλλά και προτεραιότητα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχει τεθεί από τους αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων ε, το τέλος του 2015 ως ε, προθεσμία και μετά μπορούμε να περάσουμε στην επίσημη υιοθέτηση κάποια στιγμή στις αρχές του 2016. Και μετά από δύο χρόνια φάσης υλοποίησης να έχουμε τελικά ευρωπαϊκό δίκαιο προστασία δεδομένων, το οποίο να είναι εφαρμοστέο κάποια ε, στιγμή στι αρχέ του 2018. Έχουμε βεβαίω και διαδικασίε διαβούλευση που ξεκίνησαν το 2010, αλλά τελικά θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και πραγματικά ελπίζω τα πρότυπα στα οποία θα καταλήξουμε να μην είναι κατώτερα της οδηγίας του 1995, αλλά σε ορισμένα ζητήματα να είναι και πιο ακριβή, να δίνουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και να διευκολύνουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τι εντολέ του Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσει. Βεβαίω δεν υπάρχει και χρόνο, επομένω μπορεί να γίνει διμερό στη συνέχεια. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μέχρι τι 6 και 10 ο κύριο Κύρκο δεν... δεν είναι εδώ. Παρακαλώ, Μαριόν. Ευχαριστώ Κλοντ και ευχαριστώ και το Γιάννη γιατί με διευκόλυνε, θα είναι πιο σύντομη η παρουσίασή μου. Είμαστε βέβαιοι ότι εργαζόμαστε και οι δύο προς την ίδια κατεύθυνση γιατί θέλουμε να καταλήξουμε σε τελική συμφωνία ε, μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης, έχουμε δύο τριμερείς διάλογους ακόμα και έχουμε ήδη μία πρώτη συμφωνία με το κεφάλαιο 1, χωρίς το πεδίο εφαρμογή βέβαια, το πεδίο εφαρμογή συζητιέται ακόμα, και τα κεφάλαια 3, 4, 5, 8, 9 και 10. Και τη Δευτέρα θα γίνει ο επόμενος τριμερής διάλογος, στον οποίο θα συζητήσουμε τα κεφάλαια 2, 6, 7 και 8α όπερ και σημαίνει ότι στο Στρασβούργο θα γίνει η τελευταία συζήτηση όπου θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με, ε, για τα εκκρεμή ζητήματα. Ένα από αυτά το ανέφερα, είναι το πεδίο εφαρμογή που θα πρέπει μαζί με τον κανονισμό να υπάρξει μια συνεννόηση για το πώς μπορούμε πραγματικά να ε, καλύψουμε την επιθυμία και τη ζήτηση, ο κανονισμός να καλύπτει και την ανταλλαγή δεδομένων που αφορά τον τομέα της δημόσιας ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα έχοντας κατά νου και το γεγονός ότι η δημόσια ασφάλεια είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ένας ορισμός ο οποίος ε, θα καλύπτει και το κοινοτικό δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα και τις ανάγκες των κρατών μελών. Ε, προσπαθούμε να βρούμε μια λύση γι' αυτό. Τώρα, ποια άλλα θέματα συζητιώνται ακόμα. Νομίζω ότι ένα από τα ζητήματα τα οποία ε, συζητούμε αφορά και τη Europol, είναι η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες με την ελπίδα ότι τα κράτη-μέλα σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις θα μπορούν να επιτρέπουν και την ανταλλαγή δεδομένων για ιδιωτικούς φορείς, αλλά εδώ είναι πάρα πολύ ε, σκληρές οι συζητήσεις, διότι ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε κάποια λύση. Καταρχήν ε, δεν είμαστε και τόσο ικανοποιημένοι ε, για, με το γεγονός αυτό. Προσπαθούμε λίγο να το περιορίσουμε και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Τώρα, ένα από τα ουσιαστικά ζητήματα είναι το γεγονός ότι μέχρι τώρα οι αρχέ επιβολή του νόμου δεν είχαν δυνατότητα εναρμόνιση. Είναι 28 διαφορετικές παραδόσεις, 28 διαφορετικών κρατών μελών, διαφορετικές ε, διαδικασίες και νοοτροπία ερευνών και γι' αυτό ακριβώ υπήρχαν και πολλές αμφιβολίες και φόβος μεταξύ των ε, ε, αρμοδίων του κλάδου ότι μπορεί να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά την καθημερινή τους δουλειά. Και επειδή εγώ δεν συμμετούχα μεν στην προηγούμενη θητεία, αλλά τότε επικρίθηκε ιδιαιτέρως ο διευθυντή και μάλιστα δεν πέρασε και ομόφωνα το ζήτημα λόγω των φόβων αυτών των υπολείπων. Προσπαθούμε λοιπόν με το Συμβούλιο να υπάρχει μια αμοιβαία συνεννόηση. Να γίνει κατανοητό ότι η οδηγία βοηθά να γίνεται καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύουμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων. Ε, και η αστυνομία και οι αρχές επιβολής του νόμου και οι επαγγελματίες ε, να έχουν και το ελεύθερο να μπορούν να προσαρμοστούν στην ομοτροπία τους, ε, στις επαγγελματικές τους ανάγκες και να έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν κάποια θέματα τα οποία είναι υπό έρευνα χωρίς να υπάρχει ο φόβος ότι θα υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση περιττή. Και εδώ νομίζω ότι το να αντιληφθούμε ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος του συστήματος προστασίας δεδομένων και του ε, υπεύθυνου προστασίας δεδομένων. Στη διάρκεια αυτού του τριμερούς διαλόγου ε, υπάρχει ένα και μεγαλύτερη προσέγγιση και βλέπουμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση η συνεργασία με το Συμβούλιο ήταν πάρα πολύ καρποφόρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν το Συμβούλιο που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, παρουσιάζει όλες μας τις θέσεις στα κράτη-μέλη και την τελευταία φορά, στην αρχή του τριμερής διαλόγου, υπήρξε μια σαφέστατη δήλωση ότι τώρα και τα 28 κράτη-μέλη ενδιαφέρονται να ολοκληρωθεί η οδηγία ώστε πραγματικά να ενισχυνθεί η συνεργασία και να βοηθήσει το έργο τους. Το λέω αυτό γιατί υπήρχαν κάποια πράγματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο έχουμε ένα πάρα πολύ στεναρωμένο μήνυμα ότι τα κράτη-μέλη περιμένουν να υπάρξει μια λύση. Ελπίζουμε λοιπόν να καταλήξουμε σε αυτή την αμοιβαία επωφελή λύση για του, στη διάρκεια των επόμενων δύο συναντήσεων. Είμαι βέβαιοι ότι το τελικό κείμενο θα προσφέρει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και ταυτόχρονα θα επιτρέπει και στην αστυνομία να κάνει την πολύ δύσκολη και περίπλοκη δουλειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα είναι έτοιμη η δέσμη μέτρων για την προστασία δεδομένων πριν από τα τέλη του έτους και όπως είπαμε και στο προηγούμενο θέμα σχετίζεται και με τα όλα όσα αφορούν τα στοιχεία επιβατών, το PNR. Θα υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα το οποίο πραγματικά θα μπορούμε να εφαρμόσουμε και το οποίο θα προσφέρει καλύτερες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο για την ε, πολύ ε, έκτενη παρουσίαση των δύο σημαντικών αυτών θέματων. Έχουμε δύο σκιώτες για τα θέματα αυτά. Καταρχάς ο κύριος Φως να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ο ίδιος και τα δύο θέματα. Θα ήθελα να πω λοιπόν ε, δύο πράγματα για αυτό που αποφασίσαμε πριν από δύο χρόνια. Ε, έχει βελτιωθεί κάπως το κείμενο και αυτό μου δείχνει, μου δίνει πολλές ελπίδες. Αυτό που θα ήθελα να έχει συμβεί εν τω μεταξύ, ιδιαίτερως μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, θα ήταν να είχαμε κάτι και να είχαμε ελέγξει λίγο κατά πόσον το μέσο αυτό το οποίο δημιουργούμε αποτελεί νομική βάση και για τέτοιες ε, ακραίες ε, περιπτώσεις και για τέτοιες κατεπίγουσες περιπτώσεις. Αυτό θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά την οδηγία θα ήταν κάτι επιθυμητό. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό θα ήθελα να πω το εξή. Πέρα από το γεγονός ότι έχουμε κάποιο χρονικό περιθώριο, θα πρέπει να ελέγξουμε και το περιεχόμενο. Εδώ λοιπόν πάλι αποτυπώνεται μία κατάσταση πριν από 1,5-2 χρόνια. Δεν είναι επίκαιρο λοιπόν αυτό. Και γι' αυτό πιστεύω λοιπόν το έγγραφο αυτό αποτελεί και μια χαμένη ευκαιρία αν θέλετε. Δεν θα υπάρξει πλήρης εναρμόνιση 100% και αυτό πολύ απλά γιατί θα υπάρχουν ε, ε, πολλές ε, ανοίγματο. και δεν θα έχουμε μια λύση η οποία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσει της εποχής, ε, στα μοντέλα τα οποία υπάρχουν ούτε από πλευράς ταχύτητας ούτε από πλευράς πεδίου εφαρμογής ε, θα είμαστε επίκαιροι. Θα ήθελα λοιπόν μια πιο ε, θετική αντιμετώπιση για τα ανωνυμημένα στοιχεία και για άλλα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει για το πόσο η διαδικασία χρήσης δεδομένων, όχι η μετακίνηση των δεδομένων, αλλά η διαδικασία χρήσης των δεδομένων θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Θεωρώ ότι θα χρειαζόμασταν πιο πολλά κίνητρα για να έχουμε τέτοια χρήση των στοιχείων και των δεδομένων και προκειμένου να υπάρχουν υπεύθυνοι προστασία των δεδομένων. Η προσέγγιση ανάλογα με τον κίνδυνο θεωρώ ότι είναι περιορισμένη στην εφαρμογή της. Θα έπρεπε να έχουμε πιο εκτενή εφαρμογή για να καταπολεμήσουμε την γραφειοκρατία. Και αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 76 και 77 όπως έχει το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να παραμείνουν και οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις θα πρέπει να βελτιωθούν θεωρώ και συνολικά λοιπόν πιστεύω ότι δεν θα εξασφαλίσουμε την ιδιωτική σφαίρα των πολιτών μας, ούτε θα καταφέρουμε η ευρωπαϊκή οικονομία να είναι σε μια κατάσταση που τελικά να εξισωθεί με τις επιχειρήσεις άλλων τρίτων χωρών. Άρα, ως εκ τούτου, αν είναι δυνατόν, Θα ήθελα όλα αυτά να ληφθούν υπόψη στους τρομερείς διαλόγους. Ε, περιμένω ανοιχτό πνεύμα. Θα ήθελα να σας πω ότι στο διαδίκτυο υπάρχει ήδη ένα ενοποιημένο κείμενο του Συμβουλίου για τον Βασικό Κανονισμό και θα ήθελα να παρακαλέσω ενδεχομένω τον εισηγητή να μας το διαβιβάσει το κείμενο αυτό. Ναι, σχόλιο εκτός μικροφώνου. Το θέμα όμως είναι γιατί δεν το έχουμε ήδη λάβει. Okay. Um, have... Ο Πρόεδρος. Μάλιστα, κοιτάξτε. Αν η Προεδρία και η Επιτροπή θα μπορούσαν να μας ε, αναφέρουν ε, τι γίνεται, ε, πολύ σύντομα η Επιτροπή αν θα θέλει να πάρει το λόγο να μας πει τι γίνεται. Από το Συμβούλιο ευχαριστώ. Κανένα πρόβλημα, Πρόεδρε. Οι δύο εισηγητέ και τους ευχαριστώ γιατί μας έδωσαν μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα τη κατάσταση του φορά του θερμερού διαλόγου. Επιβεβαιώνω μόνο από πλευρά Συμβουλίου ότι και από τη δική μας πλευρά θεωρούμε ότι οι διαπραγματεύσει ε, κινούνται ε, πολύ παραγωγικά για το σύνολο του πακέτου και ευχαριστώ τους ε, εισηγητέ, τους κοιόδης και όλες, και όλους τους συνεργάτες τους για την εξαιρετική αυτή δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι τώρα μπαίνουμε σε μία αποφασιστική φάση ε, των διαπραγματεύσεων. Αυτές οι επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες θα είναι κρίσιμες σημασία. Το Συμβούλιο, η Προεδρία, όλα τα κράτη-μέλη πραγματικά επιθυμούν την οριστικοποίηση της μεταρρύθμισης μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Όπως ε, αναφέρθηκε Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σε πολύ υψηλό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι επιθυμούμε την ολοκλήρωση των πραγματεύσεων μέχρι τα τέλη τη χρονιά. Και σε ό,τι αφορά την οδηγία, θα ήθελα να πω ότι και οι υπουργοί το επεσήμαναν κατά τη διάρκεια του έκτακτου Συμβουλίου Τζάι, που έγινε στις 20 Νοεμβρίου, ότι αν κατέστη κάτι σαφέ τι τελευταίε εβδομάδε, είναι ακριβώ αυτή η αναγκαιότητα ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών αρχών και δικαστικών αρχών. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε έναν αρμονισμένο πλαίσιο προστασίας δεδομένων το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει λοιπόν σαφή δέσμευση από πλευρά μα για να ολοκληρώσουμε αυτή τη μεταρρύθμιση το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε. Δεν μένει πολλή χρόνο μέχρι να περάσουμε στη ψηφοφορία και άλλοι συναδέλφοι έχουν στο λόγο. Όμω πρέπει να κλείσει εδώ με τον. Ο κύριο, η κυρία Φελτ. Δεν νομίζω ότι έχουμε χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα πολύ σύντομο σχόλιο για ένα λεπτό. Συγγνώμη για την πίεση χρόνου. 30 λεπτά λέει η ομιλήτρια. 30 δευτερόλεπτα φαντάζομαι να είτε. Η Προεδρία του Συμβουλίου με έχει διευκολύνει. Συμφωνώ με το όσο αναφέρθηκε. Να πω μόνο ότι η μεταρρύθμιση στην προστασία δεδομένων είναι από τι ε, κύριε προτεραιότητε ε, του Πρόεδρου Γιούγκερ και του συνόλου του Σώματο των Επιτρόπων. Ε, στηρίζουμε την οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων, αλλά και για την αστυνομική μεταρρύθμιση είναι κάτι πολύ σημαντικό αστυνομική συνεργασία, συγγνώμη, πολύ σημαντικό και για την καλύτερη συνεργασία των δεδομένων και για την Ευρωπαϊκή Ένωση Σε Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ιντσέλτ και μετά θα επιστρέψουμε στους συγγητές. Ναι, πολύ σύντομα. Συμφωνώ με τα όσα είπαν οι συγγητές και εγώ πιστεύω ότι κάνουμε πολύ καλή δουλειά ή μάλλον η Προεδρία του Λουξεμβούργου έκανε εξαιρετική δουλειά σε αυτούς τους δύο φακέλους όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζω να κλείσουν και οι τρεις φάκελοι, η οδηγία προς δεδομένων, κανονισμός προς δεδομένων και το PNR να κλείσουν γιατί με έχουν κουράσει <laughs> μάλιστα τόσα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερως. Έχουμε ψηφίσει την εντολή και για τους τρεις φακέλους. Μπορεί να μην μας αρέσει το αποτέλεσμα. Εμένα μου αρέσει το αποτέλεσμα σε κάποια και δεν μου αρέσει σε κάποια άλλα. Αλλά έτσι είναι η δημοκρατία. Δεν κατανοώ το ΕΛΚ και την επιμονή του ΕΛΚ που θέλει να καθυστερήσει ε, την υιοθέτηση της εντολής ε, κατά τη διάρκεια των προβετεύσεων ε, ε Εγώ θέλω να διατηρηθεί η εντολή που έχει ψηφιστεί και στη Λίμπε και στην Ορομέλεια και ελπίζω να κλείσουν αυτή η φάκελοι μέχρι λοιπόν στα τέλη της χρονιάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λόριστεν. Πολύ σύντομα για τα όσα είπε ο κύριος Φως ότι πρέπει να τα ελέγξουμε περισσότερο τα πράγματα για να καλύπτονται οι ανάγκες σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γνωρίζουμε. Όλες οι απαραίτητες ε, εξαιρέσεις που αφορούν ε, περιπτώσεις που συνδέονται με την τρομοκρατία και το καθεξής ήδη υφίστανται. Έχουν ήδη συζητηθεί και έχει υπάρξει συμφωνία. Δεν υπάρχει λοιπόν ζήτημα, πρόβλημα για το Συμβούλιο και Εκκλησιών και Συμβούλιο και εμείς ε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα πρέπει να καλύπτονται και αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστούμε Μαριού. Γιάνν, θες κάτι να πεις, κάτι τελευταίο. Ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω μόνο ότι είναι κέριο ζήτημα για την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και για την ψηφιακή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί ε, ο κανονισμό που είναι δεδομένο των μέτρα δυνατών. Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, να υπάρχει ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Ίση όρη δηλαδή, όχι μόνο για τι επιχειρήσει, αλλά και για του ε, καταναλωτέ. Πρέπει να γνωρίσουν τα δικαιώματά του στην ευρωπαϊκή αγορά. Και βεβαίω ε, να προασπίσουμε και το θεμελιώδε δικαίωμα τη προστασία δεδομένων, το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται με 28 διαφορετικού τρόπου. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε ούτε μία μέρα παραπάνω. Πρέπει να το υιοθετήσουμε αυτό πάρα αυτά και να μην καθυστερούμε και επιμηκύνουμε διαπραγματεύσει που είναι προφανές ότι ε, είναι πολύ κοντά στην ολοκληρωσή τους. Επίσης να υπενθυμίσω ότι η εντολή του Κοινοβουλίου για τον κανονισμό υπερψηφίστηκε κατά 95% από την Ολομέλεια. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα θα πρέπει να προχωρήσουμε με βάση και τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, το σημότερο δυνατόν. Η Προεδρία εργάζεται πολύ σκληρά μαζί με εμά, ε, το αναγνωρίζω, καθώς και την βούληση των 28 ε, κρατών μελών να καταλήξουμε συμφωνία. Κρεμούν κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν, όμως σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αναφέρθηκαν και από τους ευκαιώδεις που πήραν το λόγο, πρέπει να πω ότι κατά τη γνώμη μου έχουμε ολοκληρώσει την αποστολή μας και για την εισαγωγή νέων εξελίξεων και καινοτομιών στον τομέα της προσθέσεως και με την ψευδονιμοποίηση που ήταν δική μου πρόταση και ελήφθη υπόψη σε όλες τις πραγματεύσεις και αποτελεί τμήμα του πακέτου που εξετάσαμε. Αλλά και σε ό,τι αφορά την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο που έγινε κατόπιν δικής μας πρότασης του Κοινοβουλίου, τη δέχτηκε το Συμβούλιο και τώρα κινούμαστε πιο κοντά, εξετάζουμε δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει αυτή η προσέγγιση βάσει του κινδύνου στην πράξη, όμως υπάρχει μία σαφής ε, βάση με αιτήματα που έχουν ληφθεί υπόψη από όλες τις πλευρές και έχουν υποβληθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και νομίζω ότι πρέπει και εμείς να μεριμνήσουμε ή μάλλον να αναγνωρίσουμε ότι αυτές οι πραγματεύσεις ε, έγιναν με πολύ εμπεριστατωμένο τρόπο και πρέπει να γίνουν, το αποτέλεσμά τους να γίνει δεκτό και ελπίζουμε να γίνει αυτό μέσα στις επόμενες δύο συναντήσεις τριμερούς διαλόγου. Ευχαριστώ. Μια τελευταία λέξη είπα να πεις, αλλά εντάξει, δεν σε κατηγορώ. Συνάδελφοι, παρακαλώ, θα θέλετε να ψηφίσετε, σας παρακαλώ. Ε, ευχαριστούμε τους ε, σκιώτες και τους εισηγητές και τους υπόλοιπα μέλη που εμπλέκονται. Ευχαριστούμε και την Προεδρία και την Επιτροπή 10 και 15 Δεκεμβρίου επόμενη λοιπόν, τρίμερη διάλογη για την οδηγία ΔΕ στις 7 και 17 Δεκεμβρίου. Να κάνουμε διάλειμμα. Όχι, δεν κάνουμε διάλειμμα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε πάρα αυτά τις ψηφοφορίες.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 Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ, σας παρακαλώ καθίστε. Για να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, παρακαλώ. First Προς μία νομοθετική πράξη για την ενιαία ψηφιακή αγορά, Μίκαλ Μπόνι, ο εισηγητής, δεν ξέρω αν θέλει να πάρει το λόγο, αλλά εν συντομία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιότες, συζητητές, όλους τους εμπειρογνώμονες, τους συμβούλους, τους υπαλλήλους, γιατί ξεκινήσαμε την κατάρτιση της γνωματότησης. 120 ήταν οι τροπολογίες που λάβαμε και τώρα έχουμε πλέον 13 συμβαστικέ προτάσεις, κάποιες ξεχωριστές ψηφοφορίες. Ελπίζω λοιπόν ότι να αποτυπώνεται έτσι η άποψη της ΛΥΜΠΕ για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να περάσουμε πάρα αυτά στη ψηφοφορία. Συμβαστική 1. Έναρξη ψηφοφορίας, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Τώρα ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, αν ψήφισατε όλοι, ο Πρόεδρος. Εγκρίνεται η 34 ως προσθήκη ψηφίζεται έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Έναξη ψηφοφορία. Α, συγγνώμη, η 51. Η 51 ως προσθήκη. Έναξη ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Έναρξη ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρασε. Συμβαστική 8. Εγκρίνεται η 7. Συμβαστική 8. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 467. Ως προσθέκη. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Ένα ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Ένα ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Έναρξη ψηφοφορίας. Σας αφήνω λίγο παραπάνω χρόνο γιατί υπάρχει μια σύγχυση σήμερα. Ό,τι θέλετε βέβαια. Πέρασε εγκρίνεται. Συμβαστική 12, έναρξη ψηφοφορίας. Η συμβαστική 13, Αντιρθώνει ο Πρόεδρος, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο. Έναρξη ψηφοφορίας, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Συνάδελφοι, η επόμενη ψηφοφορία είναι για την στρατηγική συνεργασία για την καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκληματικότητα και τη τρομοκρατία μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και τη Ευρωπόλ. Αλεξάνδρα Μουσολίνη, συγγετρία. Να ξεκινήσουμε με την τροπολογία 1. Την 1, 2 και 3 ψηφίζουμε μαζί. Με ονομαστική κλίση. Έναρξη ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τέσσερα και 5. Ταυτόσημες. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 10. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Έναρξε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγητρία, την κυρία Μουσολινή. Επόμενη ψηφοφορία για το σχέδιο απόφασης ε, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Europol, για τη συνεργασία στη Βοσνία, Ζεργοβίνη και την Ευρωπόλ. Ο Λορέντσο Φοντάνα είναι εισηγητής. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να ψηφίσουν, επιτρέπεται πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε τώρα στην ετήσια έκθεση σχετικά με την ε, προστασία των οικονομικών σφαιρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της καταπολέμησης της απάτης. Συντάκτης της γνωμοδότησης ο Πίτερ Γιάζεκ. Περνάμε στην τροπολογία 8, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη. Το ΕΛΚ έχει έναν επιπλέον ε, που ψηφίζει. Παρακαλώ λοιπόν πρέπει να ξαναγίνει η ψηφοφορία με ένα λιγότερο. Το ξέρω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά από τεχνική σκοπιά πρέπει να είμαστε σωστοί. Να ξαναψηφίσουμε τη 13. Ένα από το ΕΛΚ παρακαλώ να μην ψηφίσει. Παράγραφο 1, τροπολογία 13. Επαναλαμβάνεται, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία 4, άρχεται ψηφοφορία, πρώτο τμήμα. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. βασικη τροπολογία 6. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30, πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορια Εγκρίνεται. Τροπολογία 30, δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Αιτιολογική σκέψη και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Πρώτο τμήμα. Πέρας ψηφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 5, δεύτερο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και με το κείμενο ως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ήταν μονομαστική κλίση η ψηφοφορία αυτή. Ψηφίζουμε το κείμενο ως τροποποιήθηκε ονομαστικά. Ήταν η τελευταία ψηφοφορία αυτή. Ζητώ συγγνώμη να διευκρινίσω ότι ήταν η τελική ψηφοφορία η οποία γίνεται με ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε λοιπόν ονομαστικά. Θέλετε να ξαναγίνει ή είστε ικανοποιημένοι. Εντάξει. Πέρασε τη ψηφοφορία. Να διευκρινίσω και πάλι ότι ήταν η τελευταία ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια στον κύριο Γέζικ. εκτείνει τη γνωμοδότηση. Λοιπόν, μία ψηφοφορία για τις προϋποθέσεις ε, των διαπραγματεύσεων εν ώψη και της ε, δεύτερης, ε, της συμφωνίας συγγνώμη, σε δεύτερη ανάγνωση. Πρόταση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τι προποθέσει εισόδου και διαμονή υπηκών τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, σπουδέ την ανταλλαγή μαθητών, την έμιση, άμυστη πρακτική άσκηση, την εθελοντική εργασία και την απασχόληση εσωτερικών άμυστων βοηθών. Η συγγήτρια είναι η κυρία Σεσίλια Βίπστρον και ε, ψηφίζουμε το κείμενο το οποίο συμφωνήθηκε στι διοργανικέ διαπραγματεύσει. Θέλει να πει η συγγήτρια κάτι? Όχι, ωραία, ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 49 ψήφοι υπέρ, 3 κατά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Another final vote. Ακόμα μια τελική ψηφοφορία σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των ε, διοργανικών διαπραγματεύσεων ε, για τον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Επιβολής του Νόμου, συνεργασία και κατάρτιση Europol, με ανάκληση αποφάσεων 2009-371, 2005-681. Αγουστίν Δίας Δεμέρα, ο εισηγητής. Παρακαλώ, θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. πάνω από 80 συνεδριάσεις και πλέον έχουμε φτάσει στη δεύτερη ανάγνωση. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ευχαριστώ πολύ στους κοιόδης εισηγητές, ε, στους συνεργάτες και τους συμβούλου τους. στο Συμβούλιο Τζάι, στο Συμβούλιο για την τόσο επικοδομητική του στάση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τόσο επικοδομητική τους ε, βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Δία μέρα. Να περάσουμε τώρα στην ε, ψήφιση του κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 43 υπέρ, 5 κατά, 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Τέλος ε, των συμφοριών.